Bien. Je vous remercie de prendre place. Είστε παρακαλώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, και αναφέρομαι βέβαια και στους συμβούλους των πολιτικών ομάδων, σας καλωσορίζω στην συνεδρίασή μας, τη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το σχέδιο πρακτικών των συνεδριάσεων της 21ης Οκτωβρίου, καθώς επίσης και της 4ης και 5ης Νοεμβρίου, είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο και σας έχουν διανεμηθεί επίσης. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, τότε μπορούμε να θεωρήσουμε ότι τα πρακτικά αυτά εγκρίνονται και μπορούμε θεωρώ να εγκρίνουμε και το σχέδιο μερίσιας διάταξης. Θα ήθελα να σας πω ότι ε, χθες ε, είχαμε την ε, δεύτερη ημέρα από τότε που ανέλαβε η νέα Επίτροπος Περιφερειακής Ανάπτυξης, η Ελίζα Φερέιρα, που ξέρετε ότι είχε περάσει από ακρόαση εδώ στην Επιτροπή μας. Εγώ τη συνάντησα από τότε που διορίστηκε και μάλιστα στενοηθήκαμε να έρθει πολύ σύντομα ενώπιον της Επιτροπής μας όσα ήθιστε. Επομένως, πολύ σύντομα θα φροντίσω να σε ενημερώσω για την ημερομηνία της συνεδρίασης αυτής, στα πλαίσια της οποίας θα μας δοθεί εκ νέου η ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις με την νέα Επίτροπο. Πρέπει να σας πω επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται επί του παρόντος ε, τις ε, τελευταίες διευθετήσεις όσον αφορά το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και η δική μας Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ε, είναι σε απόλυτη ετοιμότητα το συντομότερο δυνατό να επέμβει για τη διαμόρφωση του σημαντικότατου αυτού κανονισμού. Να επιστήσω επίσης την προσοχή σας στο ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεδριάσει σε σύνθεση ολομέλεια εκτάκτο όσον αφορά το, τη Νέα Πράσινη Συμφωνία. Πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο αφορά πάρα πολύ και τη δική μας την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης και όσο περισσότεροι τελικά είναι οι συνάδελφοι που θα είναι παρόντες στην Ολομέλεια και που θα πάρουν το λόγο για ζητήματα πολιτικής συνοχής, τόσο πιο χρήσιμη και επικοδομητική θα είναι για μας και αυτή η επερχόμενη ολομέλεια για το New Green Deal. Μπορούμε τώρα να περάσουμε στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης, όπου εδώ μετά από αίτημα της Επιτροπής μας της Ρέτζη, το θεματικό τμήμα Β ζήτησε την εκπόνηση μελέτη όσον αφορά την πολιτική συνοχή και πιο συγκεκριμένα το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τη συνθήκη τη Λισαβόνα και έπειτα. Από τότε που ετέθη σε ισχύ η συνθήκη τη Λισαβόνα, είμαστε πλέον συνομοθέτε και εμεί ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πολιτική συνοχή και επίση ώρε μπορούμε να εγκρίνουμε κανονισμούς με το Συμβούλιο όσον αφορά τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία. Επίσης, ασχολούμεθα ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με τις άτυπες διαδικασίες, όλο δηλαδή το προνομοθετικό έργο, καθώς επίσης και με τις διοργανικές συνομιλίες, ζήτημα το οποίο μας αφορά όλους ιδιαιτέρως, γιατί όπως ξέρετε, επί του παρόντος έχουμε ξεκινήσει μία σειρά από τριμερείς διαλόγους, για πάρα πολλά ζητήματα, για το ΦΕΤΕΡ, το, Ιντερεγ, για το Ταμείο Συνοχής, για τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων και ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό πάντα να τηρούν τις βασικές αρχές της συναπόφασης και ιδίω ε, όσον αφορά την ε, μέθοδο που είχε οθετήσει το Συμβούλιο για το διαπραγματευτικό πλαίσιο, το περίφημο negotiating box, το οποίο θα μπορέσουμε να συζητήσουμε και αργότερα. Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να δούμε ποιο είναι ο ρόλο και ω προ τον έλεγχο πασκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου για την πολιτική συνοχή. Η μελέτη διανεμήθηκε στα μέλη τη Επιτροπή μα ήδη από τον Ιούλιο του 2019 και θα μα παρουσιαστεί σήμερα το απόγευμα από τον κύριο Χάρη Μαρτίνο και από τον κύριο Σεραφίν Πάζο Βιντάλα. Έχουμε περίπου 45 με 50 λεπτά στη διάθεσή μας για αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης. Θα ήθελα να ζητήσω λοιπόν από τους προσκεκλημένους μας να τηρήσουν αυτό το χρόνο αγόρευσης, δηλαδή να μιλήσουν περίπου 15 με 20 λεπτά συνολικά, προκειμένου στη συνέχεια να μπορούν να πάρουν το λόγο και οι βουλευτές για να κάνουν παρατηρήσεις ή να θέσουν ενδεχόμενες ερωτήσεις. Έχετε το λόγο λοιπόν για την παρουσίαση της μελέτης σας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα σας παρουσιάσουμε τα βασικότερα σημεία της μελέτης αυτής. Και όπως το είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε, η μελέτη αυτή ολοκληρώθηκε στις αρχές Ιουλίου. Επομένως, ε, ήταν ε, στο τέλος της ε, προηγούμενης θητείας, μετά το τέλος μάλλον της προηγούμενης ε, θητείας του Κοινοβουλίου. Θα κάνουμε μια σύντομη εισαγωγή και θα δούμε τα πιο συγκεκριμένα το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις ε, πιο έντονες νομοθετικές ε, περιόδους, δηλαδή την νομοθετική δέσμη 2014-2020, την τρέχουσα νομοθετική περίοδο και θα δούμε και το ενδιάμεσο αυτό διάστημα, όπου θα δούμε τον συνεχιζόμενο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανάμεσα σε αυτές τις δύο νομοθετικές περιόδους εχ και θα καταλήξουμε έπειτα σε κάποια συμπεράσματα, σε κάποιε συστάσεις και κάποια σημεία προς περαιτέρω προβληματισμό για τις προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουμε τώρα και που θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον, που θα αντιμετωπίσει μάλλον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής. Όπως το είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε, η μελέτη αυτή εξέτασε και τις τυπικές, επίσημες και τις άτυπες διαδικασίες και εμείς αποπειραθήκαμε να κάνουμε εδώ πέρα μια κριτική ανάλυση για το ποιες είναι οι διαδικασίες αυτές, αλλά και ποια είναι τα αποτελέσματα αυτά, αυτών των διαδικασιών, τα αποτελέσματα δηλαδή πολιτικής και ποιοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι περιορίζουν τελικά αυτά τα αποτελέσματα πολιτικής. Στα πλαίσια της νομοθετικής δέσμης για την περίοδο 2014-2020, δηλαδή στην ε, τρέχουσα αυτή νομοθετική περίοδο και μέχρι το 2013, είδαμε ότι ε, μολονότι τότε είχαμε την πρώτη νομοθετική δέσμη κατά τη διάρκεια της οποίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε πλήρεις αρμοδιότητες ε, συνομοθέτη, ήδη τότε ήταν ε, σαφής η συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τότε ήταν κυρίως να προωθήσει πολλές σημαντικές πτυχές της πολιτικής συνοχής, όπως η στρατηγική προσέγγιση και ο προγραμματισμός, η αρχή της εταιρική σχέσης, η θεματική συγκέντρωση, καθώς επίσης και το κοινό στρατηγικό πλαίσιο, η ολοκληρωμένη εδαφική προσέγγιση με τις διάφορες πτυχές της, η υποστήριξη των, ε, των περιφερειών μετάβασης, καθώς επίσης και η πρόθεση της ευφυούς εξειδίκευσης. Παρ' όλα αυτά υπήρχαν και κάποιοι τομείς στους οποίους ε, οι απόπειρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να επηρεάσει τα αποτελέσματα δεν εστέφθησαν με επιτυχία. Και αναφέρομαι εδώ πέρα στην μακροοικονομική αιρεσιμότητα, στο πλαίσιο επιδόσεων, καθώς επίσης και μία σειρά χρηματοοικονομικών θεμάτων. Εν γέννη πάντως μπορούμε να πούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατάφερε μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μετά την έγκριση της συνθήκης της Λισαβόνας να αρχίσει να ασκεί τον πλήρη ρόλο του ως συνομοθέτη. Η περίοδος αυτή ήταν ιδιαίτερα έντονη, γίνανε πάρα πολλές διαπραγματεύσεις, πρωτόγνωρες πραγματικά για τον τομέα της πολιτικής συνοχής και οι διαπραγματεύσεις αυτές οδήγησαν σε πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Και κυρίως θα έλεγα ότι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν καθοριστικός στην επιβεβαίωση και την ενίσχυση των ε, χαρακτηριστικών της πολιτικής συνοχής προκειμένου να γίνει μια ολοκληρωμένη πολυτομεακή πολιτική καθώς επίσης και μια πραγματική επενδυτική πολιτική για όλες τις περιφέρειες της Ένωσης. Αναφερόμαστε βέβαια σε μια νομοθετική περίοδο όπου υπήρχε μία πολύ στενή ευθυγράμμιση ανάμεσα στις θέσεις του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό φάνηκε άλλωστε και στις διαπραγματεύσεις. Και στη μελέτη μας μάλιστα λέγεται ότι υπήρχε και ένας αποτελεσματικός εσωτερικός συντονισμός στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίω στην τότε υφιστάμενη ομάδα εργασία για την πολιτική συνοχή, που συνέβαλε πάρα πολύ στο να συντονιστούν οι προσπάθειες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στη συνέχεια ακολούθησε μία περίοδος την οποία εμείς ονομάζουμε ως η συνεχιζόμενη νομοθετική διαδικασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά την ιδιαίτερα φρενήρη αυτή περίοδο διαπραγματεύσεων ακολούθησε μία περίοδος σποραδικής νομοθετικής δραστηριότητος που εκτείνεται από τα τέλη του 2013 μέχρι περίπου το 2017. Περίοδος που ουσιαστικά ανταποκρίνεται στον πολιτική χαρακτήρα της πολιτικής συνοχής και εδώ πέρα ακολουθήθηκαν όλες οι νομοθετικές διαδικασίες κυρίως για να τροποποιηθούν οι υφιστάμενοι κανονισμοί. Παρ' όλα αυτά, ορισμένοι από τους κανονισμούς αυτούς ήταν πολύ σημαντικοί, όπως ο αποκαλούμενος κανονισμός Omnibus ο οποίος παρέτεινε περισσότερο το καθεστώς απλοποίησης για την πολιτική συνοχή. Επίσης, η δική σας Επιτροπή, η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, υιοθέτησε μια πολύ ισχυρή τοποθέτηση όσον αφορά τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα μέτρα στήριξης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, τροποποιώντας κάποια μέτρα, εγκρίνοντας ή απορρίπτοντας άλλα. Εν αντιθέσει, βέβαια, κατά τη διάρκεια της περίοδου αυτής, είδαμε ότι ήταν ε, πιο περιορισμένος ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με τον έλεγχο και την αξιολόγηση των εκτελεστικών και κατεξουσιοδότηση πράξεων. Είχαμε λιγότερες τέτοιε πράξεις οι οποίες πέρασαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όπως ξέρετε συνήθως περνούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από τις αρμόδιες επιτροπές του χωρίς πολλές τροποποιήσεις και χωρίς εκτενείς συζητήσεις. Ουσιαστικά αντικατοπτρίζεται το πέρα οι θέσει της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να αρχίσουν να εφαρμόζονται οι διατάξεις ε, του πρωτογενού δικαίου και είχαμε βέβαια και από τι διατάξει αυτές στο πλαίσιο του παράγωγου δικαίου, κατεξοδότηση και εκτελεστικές πράξεις. Θα έλεγα ότι η πιο σημαντική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της περίοδου αυτή ήταν οι εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματικά θεωρώ ότι κάλυψαν ένα πολύ μεγάλο μέρος σημαντικό θεμάτων στην πολιτική συνοχή και πραγματικά έδωσαν μια πολύ ισχυρή φωνή στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης και εν γέννη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πολιτική συνοχή. Ορισμένες από τις εκθέσεις αυτές ήταν ανταπόκριση σε σχετικές εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα έλεγα επίσης ότι ε, επέτρεψαν οι εκθέσεις αυτές στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης να ασκήσει πολιτικό έλεγχο για την πολιτική συνοχή. Ορισμένες από τις εκθέσεις αυτές ήταν ε, καθαρά νέες πρωτοβουλίες της δική σα επιτροπή και συνολικά αντιστοιχούν στα αρχικά βήματα προκειμένου να δημιουργηθεί η νέα νομοθετική δέσμη 2021-2027. Η νομοθετική λοιπόν αυτή δέσμη έχει ήδη αρχίσει να εκπονείται και θα έλεγαμε ότι είχαμε το 2017 μια πολύ σημαντική έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας όσον αφορά τους βασικούς πυλώνες της μελλοντικής πολιτικής συνοχής, έκθεση η οποία μας επέτρεψε να οριοθετήσουμε το νέο πεδίο ανάπτυξης της πολιτικής συνοχής για τη νέα περίοδο προγραμματισμού. Ε, συνέβαλε πάρα πολύ η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης η δική σας, αλλά είχατε και μια πολύ έντονη συμβολή από την ε, Επιτροπή των Περιφερειών, καθώς επίσης και από άλλους αρμόδιους ε, φορείς. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο άρχισε πάλι να λειτουργεί πλήρω ω ενωμοθέτη, θέλοντα να προωθήσει μια καλά χρηματοδοτούμενη πολιτική συνοχή και πολλές φορές αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες άρχισαν να αποκλίνουν ε, από τις αρχικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Συμβουλίου όσον αφορά την αρχή της εταιρική σχέσης για παράδειγμα ή όσον αφορά το Ταμείο για την, ε, ανάπτυξη, ε, για την Περιφερειακή Ανάπτυξη. Όπως καταλαβαίνετε όμως, παραμένουν κάποιες σημαντικές προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα επόμενα χρόνια αυτής της νομοθετικής δέσμης ορισμένες εκ των οποίων έχουν να κάνουν και με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τις σχετικές διαπραγματεύσεις. Πρόκειται εδώ πέρα για έναν ξεχωριστό τομέα, δεν υπόκειται στην αρμοδιότητα συναπόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μάλιστα πιέζει και πάρα πολύ ο χρόνος προκειμένου να επιτευχθεί μια συμφωνία για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο μέσω των τριμερών διαλόγων προκειμένου να μην καθυστερήσουν τα νέα προγράμματα της πολιτικής συνοχής. Συνοψίζοντας λοιπόν ε, τα βασικά μου συμπεράσματα, θα έλεγα ότι είδαμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αναλάβει έναν πολύ στεναρό δυναμικό ρόλο από τότε που η συνθήκη της Λισαβόνας, χρησιμοποιώντας όλες τις νέες εξουσίες που του προσδίδει η συνθήκη της Λισαβόνας προκειμένου να προασπίσει και να προάγει νέες θέσεις πολιτικής και όλα αυτά μάλιστα σε ένα γενικότερο περιβάλλον, όπου είχαμε κάποιους περιορισμούς για το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από δύο κυρίους παράγοντες. Πρώτον, οι εξωτερικές αλλαγές που είχαμε και που τροποποίησαν την τοποθέτηση της πολιτικής συνοχής στο πλαίσιο των γενικότερων ευρωπαϊκών πολιτικών και του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου, θα έλεγα ότι αναλήφθησαν πολλές πολιτικές πρωτοβουλίες από την προηγούμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία δημιούργησε νέα εργαλεία επενδύσεων, πρόωθησε διαρθρακτικές μεταρρυθμίσεις, ασχολήθηκε με ζητήματα συντονισμού πολιτικής, που πολλές φορές παρουσιάζουν κάποιες αλληλοεπικαλύψεις και μερικές φορές έρχονται σε αντίθεση κιόλας και με τις πρωτοβουλίες ε, της πολιτικής συνοχής. Υπήρχαν και κάποιες αδυναμίες όσον αφορά τις ικανότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή την μεταξύ των Επιτροπών Συνεργασία και Συντονισμού. του δώσω το λόγο στον συνάδελφό μου, τον Σεραφίν, ο οποίο θα σα μιλήσει για τι συστάσει που θέλουμε να σα κάνουμε, θα έλεγα απλώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε και να δραματίσει ένα ευρύτερο ρόλο πέρα από την προάσπιση τη πολιτική συνοχή. Θα μπορούσε να γίνει ένα θεσμικό όργανο το οποίο θα μπορεί προδραστικά, προορατικά να θεσπίζει προτεραιότητε για την πολιτική συνοχή και θα μπορούσε να δημιουργήσει επίση και κάποιες εσωτερικές δυνατότητες συνεργασίας και συντονισμού προκειμένου να μπορεί να κινητοποιήσει αλλά ακόμα και να ηγηθεί όλης αυτής της μεγάλης κοινότητας εξωτερικών φορέων γύρω από την πολιτική συνοχής. Εν γέννη θα έλεγα ότι μέχρι τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει καταφέρει να παγιώσει την θέση του ως το θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή θέση προκειμένου να εκφράσει τις ανάγκες και τις προτεραιότητες για την οικονομική, εδαφική και κοινωνική συνοχή. Μια-δυο ακόμα συστάσεις εν συντομία για το μέλλον. Η δυνατότητα του Κοινοβουλίου περιορίζεται, να παρέμβει περιορίζεται από το κανονιστικό πλαίσιο βέβαια, αλλά μπορούμε να, ε, αρισ, να βελτιώσουμε αυτά που έχουν γίνει στο παρελθόν. Ε, η Διευθύνουσα Επιτροπή, η String Committee, μπορεί να ε, συνεισφέρει σε αυτό. Μπορεί να πείτε ότι υπάρχει κάτι τέτοιο βέβαια. Αλλά ο οριζόντιος χαρακτήρας ενδεδομένου ότι το ΦΕΝΤΕΡ έχει επιστρέψει στον κανονισμό κοινών διατάξεων είναι κάτι το οποίο, στο οποίο θα πρέπει να δώσετε περισσότερη σημασία. Ε, δεν είναι μόνο όλες οι επιτροπές που πρέπει να εμπλέκονται και το τεχνικό προσωπικό. Θα πρέπει να συστηματοποιήσετε περισσότερο την συμβολή των ακαδημαϊκών, των εμπειρογνωμόνων, της ε, διεθνούς κοινότητας, δηλαδή των ανθρώπων που ασχολούνται με την ε, περιφερειακή πολιτική. Θα πρέπει να είμαστε πιο, πιο ορατικοί όταν ε, στις δράσεις μας, όχι απλώς να περιμένουμε τα πράγματα να ξέρουν και μετά να αντιδρούμε. Το Κοινοβούλιο έδειξε ηγετική στάση με τις ε, εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας, με τις ε, προπαρασκευαστικές δράσεις, αλλά και ε, θέματα όπως η βελτίωση των δεδομένων στα οποία βασίζεται το Κοινοβούλιο, των πληροφοριών δηλαδή που λαμβάνει, από ανεξάρτητες αρχές, από ανεξάρτητες πηγές, ε, πηγές διαφορετικές από τη Eurostat και της Κομισιόν, αυτό θα βοηθούσε για να ενισχύσει την θέση του Κοινοβουλίου, ιδιαίτερα στους τριμερείς διαλόγους. Παρόλο ότι η συνεργασία παραδοσιακά γινόταν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ίσω υπάρχει μια ευκαιρία να εγκαθιδευτεί, να μια συνεργασία και με το Συμβούλιο. Υπάρχει μια επιτροπή μέσα στο Συμβούλιο, η οποία ασχολείται με το θέμα της περιφερειακής πολιτικής, με την οποία ενδεχομένως θα μπορούσε να συνεργαστεί το Κοινοβούλιο. Με αυτόν τον τρόπο θα διευκολυνόντουσαν οι διαπραγματεύσει. Ίσως. Τέλο, το θέμα δεν είναι μόνο να έχουμε περισσότερα στοιχεία ή δεδομένα. Ήδη έχουν, έχει γίνει μεγάλη πρόοδος πάνω σε αυτό. Αλλά Ξέρω μάλιστα ότι και οι ακαδημαϊκοί ερευνητέ χρησιμοποιούν ε, τις δικές σας εκθέσεις, τις εκθέσεις επιτροπής σας, ε, τόσο τεκμηριωμένες είναι. Αλλά ε, υπάρχει και το θέμα της ε, προβολής του έργου, του έργου σας. τώρα που πλησιάζουμε στην διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Ίσως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να οργανώσει δράσεις, όχι μόνο εδώ, αλλά και στα κράτη-μέλη, για να προβάλλει το δικό του έργο. Τέλος, για το μέλλον τι άλλο μπορώ να πω. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επηρεάζεται από το συνολικό παρόραμα. Υπάρχει μια καινούργια Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε μια γενική ιδέα για το τι μπορούμε να περιμένουμε από αυτήν την Επιτροπή. Ίσως ε, θα πρέπει να δούμε το θέμα της πολλαπλότητας, της ποικιλία των διαφόρων οργάνων και μηχανισμών που διαθέτουμε, πώς θα επηρεάσουν αυτά ε, το μέλλον, πώς θα βελτιωθεί ο συντονισμός τους. Και επίση έχουμε και πολλές προτεραιότητες, οι οποίες πολύ συχνά έρχονται σε αντίθεση μία με την άλλη, ε, και όλες διεκδικούν χρηματοδότηση. Θα πρέπει το Κοινοβούλιο ενδεχομένω να εγγυηθεί ότι θα υποστηριχθούν αυτές οι προτεραιότητες μεν, αλλά ότι δεν θα πέσει στην ε, παγίδα να διχαστεί ε, μεταξύ αυτών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσουμε τώρα τη συζήτηση και δίνω το λόγο στην Κορίνα Κρέτου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συναδέλφοι. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο προσκεκλημένους ε, για αυτή τη μελέτη. Έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά. Θα ήθελα επίσης να επισημανώ ότι μετά από τη συνθήκη της Λισαβόνας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραματίζει βασικότατο ρόλο ως συνομοθέτης για την υιοθέτηση, για παράδειγμα, της νομοθετική δεσμής μέτρων από το 2014 έω το 2020 που έδωσε ιδιαίτερο βαρός στην πολιτική συνοχή. Έφτασε τα 750 εκατομμύρια ευρώ, αγγίζοντα όλες τις περιφερειές ε, και τους στόχους ε, ε, στρατηγικής. Ω επιτρόπο, στην ομάδα του κ. Γιούνκερ είδα από πρώτο χέρι τι ρόλο έπαιξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μέσω εκθέσεων ίδιας πρωτοβουλίας και μέσω τυπικών και άτυπων ε, εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων. Ε, αγωνίστηκε για σωστή χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής. Πολύ σημαντικό για όλες τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω όλης αυτής της δράσης, ε, πιστεύω, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βοηθά στη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Επειδή κάποιες περιφέρειες ακόμα χρειάζονται βοήθεια με βασικά πράγματα, όπως ε, διαχείριση απορριμμάτων, υδάτων, μεταφορές και το καθεξής. Άλλες χρειάζονται περισσότερη βοήθεια για την έρευνα και την καινοτομία. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι όπως είπε ο Πρόεδρος ο Μαζέ στην αρχή και όπως υπογραμμίστηκε στη μελέτη, η υιοθέτηση του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου πιστεύω επιβάλλεται. Είναι κρίσιμη σημασία ώστε να μπορέσουμε να αποφύγουμε να θέσουμε σε κίνδυνο τα πολυάριθμα ευρωπαϊκά έργα που τρέχουν όπως και τα νέα έργα που θα ξεκινήσουν. Ελπίζω λοιπόν το Κοινοβούλιο, η Κομισιόν και το Συμβούλιο να έχουν μια γαστή συνεργασία. Εκτιμώ ιδιαίτερα τη σύσταση για καλύτερη σχέση με το Συμβούλιο. Ωστόσο, αυτό θα εξαρτηθεί από τη βούληση αμφότερων των πλευρών. Διότι όπως γνωρίζουμε, χρειάζονται δύο για να χορέψουν ταγκό. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Merci beaucoup. Ευχαριστούμε πολύ. Αντρέι Ντόντεκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και τους συναδέλφους από την EPRS, λέει ο κ. Κνότεκ, για την ε, πλήρη αυτή μελέτη. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Τη διαβάσαμε με μεγάλο ενδιαφέρον και ακούσαμε με μεγάλο ενδιαφέρον πώς εξελίχθηκε ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πώς αυτό επηρεάζει τις δυνατότητες που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετέχει σε διάφορες πτυχές της πολιτικής συνοχής. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να τονίσουμε ότι υπάρχει μια συνέχεια και για τα νέα μέλη, όπως εγώ παρατηρώ ότι πολλοί όροι, πολλά εργαλεία που χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή έχουν τη ρίζα τους σε πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι πολύ καλό αυτό και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Επιπλέον, έχω μια ερώτηση για να βεβαιωθώ ότι κατάλαβα καλά τη σχέση μεταξύ των συστάσεων και των βασικών πορισμάτων, ε, απευθυνώ την ε, ερώτηση στους δύο μιλητές. Αναφέρατε ότι το Κοινοβούλιο έχει να παίξει σημαντικό ρόλο. Μεγαλύτερο ρόλο στο καθορισμό των θέματων της, του σημερισίας διάταξης, στην ατζέντα. Μιλήσατε για τους προενεργούς ε, κύκλους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Αντρέ. Κωνσταν Σκρέλ. Ναι, ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και για τη μελέτη και για τις ενδιαφέρουσες συστάσεις. Βοηθούν πολύ, πιστεύω. Έχω όμως μια ερώτηση για μία από αυτές. Κανείς δεν μπορεί να διαμαρτυρηθεί εδώ ότι δεν είχαμε επαφή με πάρα πάρα πολύ κόσμο. Γιατί λοιπόν δεν υπάρχει μια steering committee. Στις ομάδες έχουμε οριζόντιες ομάδες εργασίας που συνεργάζονται ε, μεταξύ πολλών επιτροπών, με μέλη από πολλές επιτροπές. Ε, οπότε εγώ αποκτώ την εντύπωση ότι προσπαθούμε να μειώσουμε τη γραφειοκρατία ε, και ξαφνικά λέμε ε, ε, φτιάχνουμε διάφορες steering committee και γεμίζουμε τα χρονοδιαγράμματά μας και τελικά δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε τη δουλειά πραγματικά. Ίσως δεν κατάλαβα καλά, θα μπορούσατε να με εξηγήσετε ποια είναι η προστιθέμενη αξία που θα προσέφερε μια τέτοια steering committee. Ευχαριστώ. Merci, Ευχαριστούμε Κωνσταντς. Υπάρχουν κάποια, υπάρχει κάποιος που θα ήθελε να πάρει το λόγο. Δεν βλέπω. Σας ευχαριστώ πολύ για τη μελέτη σας και για τις συστάσεις σας. Τα προβλήματα που θέτετε είναι πολύ σημαντικά. Θεωρώ ότι μετά από τη συνθήκη της Λισαβόνας σταδιακά Ε, συνθέσαμε την ομολογία της συναπόφασης. Και εμείς, ε, η Επιτροπή Ρέτζη, αλλά και ευρύτερα ολόκληρο το Κοινοβούλιο, σε γενικές γραμμές, σταθήκαμε στο ύψος των νέων αυτών ε, ευθυνών και αρμοδιοτήτων που μας καθιστούν πλήρους, πλήρης συνομοθέτες αλλά αυτή η νομολογία συνεχίζει να κατασκευάζεται και να οικοδομείται. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε στους διάφορους τριλόγους που έχουν ξεκινήσει και στο όσα κάνουμε εμείς ε, για να επιβάλλουμε τον αυστηρότατο σεβασμό της αρχής της ε, συναπόφασης. Σε αυτό το πλαίσιο η Κορίνα Κρέτου έχει απόλυτο δίκιο που το λέει οι σχέσεις που πρέπει να έχουμε με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σχέσεις οι οποίες πρώτα απ' όλα πρέπει να βασίζονται σε μία αρχή ισότητας. Εμείς είμαστε οι δημοκρατικοί αντιπρόσωποι των Ευρωπαίων πολιτών. Οι δημοκρατικοί τους εκπρόσωποι και λόγω αυτού μας του ρόλου έχουμε μία σχέση ανάλογη με το Συμβούλιο. Πρέπει να είστε βέβαιοι λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι οι πολιτικέ συζητήσει με το Συμβούλιο στο πλαίσιο, αν μη τι άλλο, των διαπραγματεύσεων, των διοργανικών διαπραγματεύσεων, θα πρέπει να είναι διαρκής και συνεχής μεταξύ όλων των εισηγητών και συνεισηγητών Και όσο πιο δύσκολες είναι οι σχέσεις, τόσο περισσότερες ε, είναι αυτές οι συνομιλίες. Ε, όσο πιο περίπλοκα είναι τα καθήκοντα. Ε, υπενθυμίσατε πλήρως το ρόλο της Επιτροπής μας για το σύνολο των νομοθετημάτων που έχουν ε, υιοθετηθεί σε θέματα συνοχής και πράγματι εμείς σταθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων και ήταν, αναφέρατε και αυτό, ήταν πολύ σημαντικό, θα θυμάστε, θα το θυμάται και η Κορίνα Κρέτου, τα ειδικά μέτρα που λάβαμε για την Ελλάδα, τα οποία λήφθησαν πάρα πολύ γρήγορα όταν χρειάστηκε. Όπου ε, αυξήσαμε τα επίπεδα συγχρηματοδότησης έως το 100% διότι ήταν πολιτικά αεπιβεβλημένο. Καταφέραμε δηλαδή να αντιδράσουμε σωστά και η πολιτική ατζέντα είναι αλήθεια πολύ συχνά προέρχεται από το Συμβούλιο ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και εκεί πράγματι πρέπει ακόμα να σημειώσουμε κάποια πρόοδο. Θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη δυνατότητα και ταχύτητα αντίδρασης και για να καθορίσουμε τη δική μας πολιτική ατζέντα. Πρόκειται για μια ευθύνη όχι μόνο της δικής μας Επιτροπής, της ε, Ρέτζη, αλλά ολόκληρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν τα πράγματα σήμερα τελικά ε, αντιδράμε σε μια πολιτική ατζέντα που αποφασίζεται εξωτερικά από άλλους. Φυσικά υπάρχουν οι εκθέσεις πρωτοβουλίας. Η κυρία Βαντερ Λάιεν όταν ήρθε ε, ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είπε ρητά ότι έχει τη βούληση να αποκριθεί στο ε, δικαίωμα πρωτοβουλίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά αυτό που έχουμε να πούμε στο εξή στην ε, κυρία Βαντερλάιν, στην πρόεδρο της Κομισιόν, είναι ότι οι εκθέσει, οι ιδέε πρωτοβουλίε που έχουν υιοθετηθεί στι διάφορε δικέ μα επιτροπέ ε, αποτελούν μια πολύ σοβαρή νομική βάση. Ειδικότερα αυτέ που έχουν υιοθετηθεί εδώ στην Επιτροπή Ρέτζι. Πολύ συχνά έχουμε αποτελέσει εμεί τη ρίζα διαφορών νομοθετημάτων. Ε, θυμηθείτε τι ε, μακροπεριφερειακέ στρατηγικέ. Αυτέ προήλθαν, έχουν τη ρίζα του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. και η έννοια των εξόχως απόκεντρων περιοχών επίσης ε, περιφερειών επίσης προέρχεται από έναν ευρωβουλευτή ο οποίος ονομαζόταν Λιζιός, ο οποίος ήταν και αυτός που υιοθέτησε τη σχετική έκθεση και οδήγησε σε αλλαγή των συνθήκων. Και στην τελευταία θητεία διάφορες ε, εκθέσεις πρωτοβουλίας που υιοθετήσαμε, τις εμπνευστήκαμε, ε, εμείς ε, και αποτέλεσαν έμπνευση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις ε, επακόλουθους, επακόλουθους κανονισμούς που ε, παρουσίασε σε εμά. Τέλος, όσον αφορά τη μόνιμη Επιτροπή και στην πραγματικότητα η ερώτηση που θέτετε εσείς είναι ο εγκάρσιος χαρακτήρας και η ανάγκη επιβολής συνοχής και συνδυασμού και ευθυγράμμισης όλων των πολιτικών. Πιστεύω ότι αυτή η ευθύνη είναι ευθύνη όλων των επιτροπών όλες οι κοινοβουλευτικές επιτροπές πρέπει να υιοθετούν ε, το στόχο αυτό της συνοχής όπως θεσπίζεται στη συνθήκη. Εμείς λοιπόν ε, θα πρέπει να δράμε στο πλαίσιο αυτών των επιτροπών ώστε να λαμβάνονται υπόψη αυτοί οι στόχοι. Αλλά αυτό το πλαίσιο υπάρχει. Έχουμε πολιτικά πλαίσια άτυπα πολύ συχνά αλλά ενδεχομένως θα χρειαστεί να βρούμε και μέσα για να τον ενισχύσουμε. Σε κάθε περίπτωση και είναι κάτι καινούριο. Όσον αφορά τις συζητήσεις μας για ε, το διευκόλυνση συνδέοντας στην Ευρώπη, Έχουμε μαζί με την Επιτροπή Προπολογισμών ένα κοινό πλαίσιο για να προχωρήσουμε μαζί στη μάχη ε, ενώπιον του Συμβουλίου και εκεί έχουμε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Συγγνώμη, στον κανονισμό περί κοινών διατάξεων. Η Επιτροπή μας λοιπόν για τις περιφερειακές υποθέσεις ε, θα είναι ανοιχτή και θα παραμείνει ανοιχτή για να ακούσει ο, τις απόψεις των τοπικών περιφερειακών φορέων και για διάφορους ε, εμπειρογνώμονες ε, και φορείς σημαντικούς σε θέματα συνοχής. Σας έχουν τεθεί ερωτήσεις. Ε, σας δίνω το λόγο για να απαντήσετε. Okay, thank you. Uh... Some of these points are... Ευχαριστώ πολύ. Όντως, ορισμένα από τα ζητήματα αυτά είναι αντιλένδετα. Επομένως, θα προσπαθήσω να απαντήσω ομαδικά στις ερωτήσεις αυτές και ενδεχομένως και ο συνάδελφος Σεραφίν θα μπορέσει να προσθέσει κάποια στοιχεία. Όντως, έχουμε έναν προδραστικό, προορατικό ρόλο. Ωστόσο, όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα ότι η θέση που υιοθετούμε είναι κάπως αμυντική. Και είναι πολύ σημαντικό να το δει αυτό η δική σας η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί υπάρχουν σημαντικές πτυχές της πολιτικής συνοχής που τίθενταν ένα αμφιβόλο και εμείς θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να υπερβείτε το στάδιο αυτό το αμυντικό και θα έπρεπε να αναλάβετε ένα ρόλο λίγο πιο προορατικό, να αρχίσετε εκ των προτέρων, να προτιμάσετε το έδαφος για τις μελλοντικές συζητήσεις και να χρησιμοποιήσετε γι' αυτό και την δημοκρατική νομοποίηση που σας δίνει με ένα πολύ πιο ισχυρό τρόπο και η ίδια η συνθήκη της Λισαβόνας θα πρέπει η δημοκρατική αυτή εκπροσώπηση να μεταφραστεί σε κάτι πολύ πιο στεναρό. Αυτό το οποίο συμβαίνει επί του παρόντος και το διακομωδώ κιόλας λίγο κάπως, είναι ότι έχουμε εκατοντάδες προτάσεων που φτάνουν από τοπικές περιφερειακές αρχές, από ενώσεις πόλεων, περνάνε μέσα από το θεσμικό ευρωπαϊκό σύστημα, χωρίς ουσιαστικά να έχουν κάποιον αντίκτυπο. Νομίζω ότι ε, το πρόβλημα είναι εδώ πέρα, ότι ε, μπορούμε να καταλήγουμε σε ένα ε, ευέλικτο μοντέλο, αλλά θα λέγαμε ότι εσείς από το να συνδυάζετε μεταξύ τους τις διαφορετικές αυτές προτάσεις και να τις συλλέγετε απλώς, θα πρέπει να τις προωθείτε και λίγο περισσότερο, να εκμεταλλεύεστε ουσιαστικά όλες αυτές τις προτάσεις που σας φτάνουν και Ανταυτού βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφιερώνει πάρα πολύ χρόνο για να αφογκράζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα προπαρασκευαστικά στάδια, προτού υποβάλει επίσημα ένα σχέδιο πρότασης. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να ακούτε ένα μήνυμα το οποίο είναι πολύ πιο συνεκτικό και η βασική ιδέα πίσω από τη θέσπιση μιας διευθύνουσας επιτροπής είναι το εξή. Ένα από του κινδύνου που αντιμετωπίζει και τώρα, αλλά και που αντιμετώπιζε και στο παρελθόν η πολιτική συνοχή, ήταν η διάσπαση σε επιμέρου τομεακέ πολιτικέ. Και υφίσταται όντω ο κίνδυνο αυτό, γιατί ακόμα βλέπουμε ότι υπάρχουν ανταγωνιστικέ μεταξύ του προτεραιότητε. Από τη φύση της, η πολιτική συνοχή ούτως ή άλλως καλύπτει τις αρμοδιότητες πολλών διαφορετικών κοινοβουλευτικών επιτροπών. Αυτό το γνωρίζετε. Επομένω, είναι πάρα πολύ σημαντικό να βασιστείτε στα δικά σας δυνατά σημεία, προκειμένου να στέλνετε προς τα έξω ένα πολύ πιο συνεκτικό μήνυμα, συγκεκριμένα προς το Συμβούλιο και δυστυχώς δεν υπάρχουν επίσημοι διάβλοι για τον διάλογο αυτό. Επικοινωνείτε με το Συμβούλιο μόνο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Και βέβαια θα πρέπει να είναι πιο συνεκτικό το μήνυμά σας και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκεί είναι πιο επίσημο, αν θέλετε, ο διάβλο επικοινωνία σα. Είναι πολύ σημαντικό τέτοιο διάβλο να θεσπίσετε όμω και με το Συμβούλιο. Γι' αυτό το λόγο σα κάνουμε τι συστάσει αυτέ, οι οποίε συνδέονται μεταξύ του και το πιο σημαντικό μα μήνυμα είναι να μην αμήνεστε απλώ των αρχικών σα τοποθετήσεων αλλά να μπορείτε να υγείστε και τη όλη διαδικασία. Τα τελευταία χρόνια είδαμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε πολλέ πρωτοβουλίε, οι οποίε ήταν πολύ σημαντικέ για την πολιτική συνοχή και οι οποίε όμω δεν μπορούσαν να ενταχθούν στο εφιστάμενο πλαίσιο αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επομένως δεν ευωδόθηκαν οι προτάσεις αυτές. Ολοκληρώνω στο σημείο αυτό. Θα ήθελα και εγώ να συμπληρώσω λίγο την απάντηση του ε, συναδέλφου μου. Να ευχαριστήσω τα όσα είπατε και τα όσα είπε και ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης όσον αφορά τις νέες ε, δομές. Αυτό το οποίο σας προτείνουμε δεν είναι να δημιουργήσετε νέα θεσμικά όργανα, νέου φορεί. Ουσιαστικά θα πρέπει να έχετε λίγο πιο συστηματικές μεθόδους εργασίας στον τρόπο με τον οποίο συλλέγετε πληροφορίες και στον τρόπο με τον οποίο απευθύνεστε σε εξωτερικούς εμπειρογνώμονε φορείς και το καθεξής. Θα υπάρχει λοιπόν κατά αυτόν τον τρόπο μια πιο συστηματοποιημένη ροή πληροφοριών που θα οδηγήσει σε μια πιο συνεκτική και στεναρή τοποθέτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την πολιτική συνοχή. Δεν σα λέω να θεσπίσετε νέε δομέ. Αρκετέ υπάρχουν άλλωστε, αλλά να έχετε ένα πιο συστηματικό τρόπο συλλογή πληροφοριών και δεδομένων και να μπορείτε να κινητοποιείτε καλύτερα την ενδιαφερόμενη αυτή επιστημονική κοινότητα. Ενδεχομένω να χρειάζεται και μια πιο διαρθρωμένη προσέγγιση, όχι μόνο για τη δική σα την Επιτροπή, αλλά παντού στο Κοινοβούλιο όσον αφορά τον έλεγχο των κατεξουσιοδότηση πράξεων. Εμεί αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή είναι ότι το υφιστάμενο σύστημα αξιολόγηση των πράξεων αυτών δεν είναι αρκετά αποτελεσματικό. Ενδεχομένω να υπάρχει στο πλαίσιο κάθε κοινοβουλευτική επιτροπή μια επιμέρου ομάδα εργασία που να μπορεί να αξιολογεί και να ελέγχει τι προτάσει αυτέ και εν τέλει να τι εγκρίνει. Αυτό αποτελεί πρόκληση όχι μόνο του δικού σα κοινοβουλίου, αλλά οποιοδήποτε κοινοβουλίου, ακόμα και των εθνικών κοινοβουλίων που καλούνται να αξιολογήσουν εξοδότηση πράξη ακόμα και για τι εθνικέ νομοθεσίε. Τα κοινοβούλια που έχουν το σύστημα αυτό που σα πρότεινα τελικά καταφέρνουν και αξιολογούν πολύ καλύτερα τι εξοδότηση πράξη. Τέλος, όσον αφορά το ζήτημα των σχέσεων που θα πρέπει να έχετε με το Συμβούλιο. Ο πρόεδρος έχει απόλυτα δίκιο όταν λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα σεβασμού και αμοιβαιότητος με το Συμβούλιο και εν τέλει ισότητος. Και προφανώς, όπως πήγε η κυρία Κρέτσου, χρειάζονται δύο για να χορέψει κανείς. Αλλά θα μπορούσαμε να είχαμε έναν πιο διαρθρωμένο διάλογο με τις προεδρίες των επιτροπών και όπως ξέρετε πολλές από τις συζητήσεις πολιτικής που γίνονται στην πολιτική συνοχής ε, γίνονται και σε εξωτερικούς φορείς, πολλές φορές ε, στα σημεία επαφής που υπάρχουν με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, με φορείς οι οποίοι είναι διακυβερνητικοί, άλλοι ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου όχι μόνο συμμετέχουν τα κράτη-μέλη, αλλά και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και άλλοι οργανισμοί μετά από πρόσκληση. Ενδεχομένως να μπορούσε και εκεί να συμμετέχει περισσότερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να υπάρχει ένα συνεχής διάλογος με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με το Συμβούλιο πέρα δηλαδή από τους επίσημους τριμερείς διαλόγους. Ξεκινάει μια νέα νομοθετική θητεία. Έχουμε ένα νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μια νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενδεχομένω να μπορούσατε να εξετάσετε λίγο αυτό με τους συνομιλητές σας, Συμβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Για μία ακόμη φορά σας ευχαριστώ για την παρουσίαση της μελέτης αυτής και για τις συστάσεις αυτές που μας απευθύνατε και επί των οποίων γύρονται κάποια ζητήματα όπως η κατεξοδότηση πράξης. Το ζήτημα αυτό είναι πολύ σημαντικό, θα μας απασχολήσει σίγουρα και θα πρέπει και με τους υπόλοιπους προέδρους των υπολείπων κοινοβουλευτικών επιτροπών να δούμε πώς θα καταφέρουμε να διευθετήσουμε το ζήτημα αυτό, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν αφορά μόνο τη δική μας την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, αλλά και όλες τις υπόλοιπες. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο της μερίσιας διάταξης. Ξέρετε ότι η Επιτροπή μας, η Ρέτζη, ανανεώθηκε πάρα πολύ. Κατά τα δύο τρίτα της, τα δύο τρίτα των μελών μας είναι νεοπλεγέντα μέλη. Τον Δεκέμβριο λοιπόν του 2014 είχαμε ορισμένες ε, ακροάσεις, ορισμένες ενημερωτικές συνεδρίες μάλλον, προκειμένου τα νέα μέλη τότε να μπορούν να έχουν μια πιο ξεκάθαρη εικόνα των ε, αρμοδιοτήτων ε, που έχουν στο πλαίσιο της Επιτροπής μας αυτής και σε σχέση βέβαια με τους συνομιλητές που έχουν από τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα. Γι' αυτό το λόγο ζητήσαμε για μια ακόμη φορά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας κάνει τρεις ε, ενημερωτικές παρουσιάσεις, ε, διάρκειες περίπου 15 λεπτών, για το ζήτημα της εξέλιξης της πολιτικής συνοχής της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το 2014, αλλά και σε σχέση με τα βασικά χαρακτηριστικά της περίοδου προγραμματισμού 2014-2020 και όσον αφορά την εφαρμογή της, καθώς επίσης και μια παρουσίαση για την πολιτική συνοχή μετά το 2020. Κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να καλύψουμε το σύνολο των ε, περιόδων αυτών προγραμματισμού θα πρέπει να μας απασχολήσουν στο πλαίσιο της τρέχουσας θητείας. Ο κύριος Έρικ Βοντράσκα, διευθυντής από την Γενική Διεύθυνση Ρέτζιο, θα κάνει τις δύο παρουσιάσεις, καθώς επίσης και ο κύριος Μωρέ Τζίλαντ, επικεφαλής μονάδας ανάπτυξης, πολιτικής ανάπτυξης, οικονομικής ανάλυσης της DG Regio. Ο κύριο Βομπρέσκα είναι παρόν από ό,τι βλέπω. Σας δίνω λοιπόν ευθύ αμέσω το λόγο για 15 λεπτά. Και έπειτα το λόγο θα πάρω στον αδελφό σα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μας καλέσατε. Θα αναφερθώ στην ιστορία της ε, πολιτικής συνοχής καταρχήν. Είναι σημαντικό αυτό για να ξέρουμε από πού ήρθαμε από που ξεκινήσαμε και που βρισκόμαστε. Πρόκειται για τη λέξη ελεγγύη, ευρωπαϊκή ελεγγύη, για να διασφαλίσουμε ότι κανένας πολίτης και καμία περιφέρεια της Ευρώπης δεν θα μείνει πίσω, δεν θα μείνει στο περιθώριο. Αυτό είναι ο στόχος της ε, πολιτικής συνοχής. και η πολιτική συνοχή ήδη βρισκόταν στη συνθήκη της Ρώμης από το 1957. Ε, ε, οι ιδρυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης το είχαν ήδη στο μυαλό τους. Βέβαια, εκείνη την εποχή δεν είχε προταθεί πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης, διότι θεωρείτο ότι το εσωτερικό εμπόριο θα οδηγούσε αυτόματα σε εναρμόνιση από μόνο του. Το πρώτο που δημιουργήθηκε ήταν το, το κοινωνικό ταμείο το οποίο υπάρχει σήμερα. Ε, δεν συνέβη βέβαια αυτό που είχαν προβλέψει οι ιδρυτές. Ε, οι διαφορές αυξήθηκαν αντί να μειωθούν. Ε, οπότε δημιουργήθηκε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης το 1975 ε, κατόπιν και της ε, πρώτης ε, διεύρυνσης της ευρωπαϊκής κοινότητας, της ΕΟΚ, με την είσοδο του Ηνωμένου Βασιλείου. Τότε δεν υπήρχαν προγράμματα, υπήρχαν μόνο σχέδια, δεν υπήρχαν δηλαδή στρατηγικοί στόχοι, δεν υπήρχαν ευρωπαϊκοί στόχοι. Μιλούσαμε για εθνικά σχέδια, πολύ απλά, τα οποία επέλεγαν τα ίδια τα κράτη-μέλη ε, με κάποια ευρωπαϊκή επίδραση, επιρροή ε, και τα χρηματοδοτούσε η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Επίσης δεν συμμετείχαν καθόλου οι περιφερειακές και τοπικές αρχές. Καταλαβαίνετε πόσο πολύ έχουν αλλάξει τα πράγματα από τότε μέχρι σήμερα. δεκαετία του 1980 με το πρόγραμμα της ε, ενιαίας αγοράς, εσωτερικής αγοράς ε, χρειάστηκε να διασφαλιστεί ότι όλοι θα υποφεληθούν από το άνοιγμα των εσωτερικών αγορών. Οπότε χρειάστηκε να δοθεί έμφαση στην περιφερειακή διάσταση η οποία αναπτύχθηκε σιγά σιγά αλλά σταθερά σε αυτό που έχουμε σήμερα. Η βασική μεταρρύθμιση είναι αυτή που περιλαμβάνει κατά βάση όλες τις ε, σημερινές αρχές της περιφερειακής πολιτικής. Ήταν αυτή που έγινε το 1988 υπό την ηγεσία του Ζακ Ντελόρ Ε, το 1988 σε αυτή τη μεταρρύθμιση λοιπόν περάσαμε στα πολιετή προγράμματα, όχι πια πλέον μόνο σχέδια, με πολιετή δημοσιονομικό προγραμματισμό, με συγκέντρωση πόρων σε συγκεκριμένους στόχους, ε, με εταιρικέ σχέσεις με τους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς και επίσης εκείνη την εποχή αυξήθηκε στο 25% του συνολικού προπολογισμού ο προπολογισμό των Ταμείων Συνοχή. Εδώ βλέπουμε τις υπόλοιπες αλλαγές που έγιναν αργότερα, μετά την μεταρρύθμιση του 1988, ε, από το τέλος δηλαδή της δεκαετίας του 80 και μετά. Από το 94 μέχρι το 99, το Ταμείο Συνοχής που εξακολουθεί να υπάρχει, ε, δημιουργήθηκε έτσι ώστε να βοηθηθούν οι, πιο φτωχές χώρες ε, να διευκολυθούν να ανοίξουν τις ε, αγορές τους χωρίς να ανατραπούν. Ε, από το 2000 στο 2006 αυτό που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι προφανώς η Ατζέντα 2000, το θεματολόγιο 2000 που προετοίμαζε την Ευρωπαϊκή Ένωση για την διεύρυνση έγινε μια προετοιμασία να ε, υποδεχθούμε τις 10, 12 και μετά 13 νέες χώρες. για την περίοδο 2007-2013 ε, να υπογραμμίσω ε, ως νεοτερισμό ότι όλες οι περιφέρειες Ευρώπης γίνονται πλέον επιλέξιμες για τα ταμείο συνοχής, όχι μόνο ορισμένε. και επίσης και κάτι άλλο, μια άλλη πρωτοτυπία, ότι η πολιτική πλέον ε, συνδέθηκε με την πολιτική της Λισαβόνας για την ανταγωνιστικότητα, όπως ονομάζεται, την στρατηγική της Λισαβόνας. Οπότε χρηματοδοτούνται επενδύσεις που θα βοηθήσουν και στην ανταγωνιστικότητα. Ε, το Ίντερεκ επίσης γίνεται στόχος, συνεργασία δηλαδή μεταξύ διαφόρων περιφερειών, και το Ίντερεγ ανήλθε πλέον στο επίπεδο των υπόλοιπων εργαλείων της πολιτικής ε, συνοχής και έγινε λοιπόν ένας ακόμα στόχος. Για την περίοδο 2014-2020 που διατρέχουμε αυτή τη στιγμή, η βασικότερη καινοτομία ήταν ότι δώσαμε περισσότερο βάρος στα αποτελέσματα και την επίδοση. Μετράμε πλέον με αρκετή ακρίβεια το τι συμβαίνει με τα χρήματα τα επενδύουμε, προκειμένου να καταλάβουμε τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί. Επίσης εισάγαμε ε, την ρεσιμότητα, ρεσιμότητα εξάντε και την μακροοικονομική ρεσιμότητα ε, που έχει σχέση με τις διαδικασίες οικονομικής διακυβέρνησης και ήταν επίμαχη ως έννοια. Τέλος, όλη μας αυτή η πολιτική συνδέεται στενά με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020. Τώρα για την περίοδο 2021-2027, θα ξανάρθω σε αυτήν την περίοδο βέβαια αργότερα, νομίζω θα συνεχίσουμε στην ίδια κατεύθυνση. Νομίζω ότι θα εστιάσουμε στην απλοποίηση και στην βιώσιμη ανάπτυξη, στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά όπως είπα θα επανέλθω σε αυτό το θέμα. Θα ήθελα να σας δείξω κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον από αριστερά προς τα δεξιά, πώς άλλαξε η επιλεξιμότητα με την παρό του χρόνου. Βλέπετε κάποια άσπρα σημεία αριστερά, ε, από το 89 στο 93, ενώ στην περίοδο 2014-2020 καλύπτονται πλέον όλες οι περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την πολιτική συνοχής. Αυτή η γεωγραφική διεύρυνση συνοδεύτηκε από μια συγκέντρωση πόρων σε ένα περιορισμένο αριθμό στόχων. Βλέπετε λοιπόν πώς εξελίχθηκε αυτή η πολιτική με το χρόνο. Τελειώνω αυτή την αναδρομή με μία-δύο διαφάνειες για το αποτέλεσμα της πολιτικής συνοχής. Έχουμε θετικό αποτέλεσμα. Εδώ βλέπετε το αποτέλεσμα της δράσης μας ε, να εκτιμήσουμε, της προσπάθειάς μας να εκτιμήσουμε πώς επηρεάζουμε ε, από το 2007 μέχρι το 2023 το ΑΕΠ, την αύξηση του ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28. Βλέπετε την μπλε γραμμή που είναι πολύ απότομη. Ξεπερνάει ακόμα και το 5%. Είναι η αύξηση του ΑΕΠ στα νέα κράτη-μέλη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη δικαιούχη των ποσών των πόρων αυτών. Βλέπετε πόσο σημαντικά έχουν αυξήσει την ανάπτυξή τους. Αλλά ταυτόχρονα θα δείτε και την πράσινη γραμμή κάτω που αφορά τις χώρες οι οποίες είναι καθαροί χρηματοδότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμα και αυτές οι χώρες έχουν έμεσες, έμεσο όφελος από την πολιτική συνοχής, γιατί, γιατί οι επιχειρήσεις τους ε, δραστηριοποιούνται στο εμπόριο με τις χώρες κεντρικής Ανατολής Ευρώπης, οπότε έχουν ε, κέρδη από αυτές τους τις συναλλαγές και κέρδη τα οποία επιστρέφουν στις χώρες που χρηματοδοτούν την, την ε, πολιτική συνοχής. Βλέπετε λοιπόν ότι και αυτή η γραμμή ανεβαίνει, έχει ανωδική πορεία. Προφανώς ε, βέβαια χαμηλότερο το όφελος αυτών των χωρών σε, σχέση με το, ως ποσοστό του ΑΕΠ σε σχέση με τις κοινέ χώρες. Λογικό αυτό. Τώρα, εδώ έχετε πιο συγκεκριμένα στοιχεία. Περίοδος 2007-2013, οι επιτυχίες μας. Συνδράμαμε περίπου 400.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δημιουργήσαμε 1,3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Συνδέσαμε περίπου 21 εκατομμύρια ανθρώπους, άτομα με νέα ευρυζωνικά δίκτυα και χτίσαμε πάνω από 6.000 χιλιόμετρα δρόμων ε, στο πλαίσιο των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Αυτά είναι πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και, και μην ξεχνάμε ότι αυτή είναι μια περίοδος στην οποία η Ευρώπη πέρασε, ζούσε μια βαθιά δημοσιονομική κρίση. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντική είναι η πολιτική συνοχής ήταν η πολιτική συνοχή τα τελευταία χρόνια. Α σταματήσω εδώ. Είναι, ήταν η πρώτη από τι τρει παρουσιάσει που έχουμε και μπορώ να απαντήσω σε ερωτήσει σα. Ευχαριστώ. Merci Σας ευχαριστούμε πολύ. Μπορούμε να προχωρήσουμε με τις παρουσιάσεις και θα ακούσουμε μετά τα σχόλια των συναδέλφων όλα μαζί και τις ερωτήσεις τους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παίρνω εγώ τον λόγο λοιπόν για το μεσό κομμάτι της παρουσίασης. Θα σας μιλήσω για τη σημερινή προγραμματική περίοδο 2014-2020. Στόχος μου είναι να σας εξηγήσω τη λογική στην οποία βασίζεται η προσέγγιση. Τι προσπαθούμε να επιτύχουμε σε αυτή την προγραμματική περίοδο στο τέλος. Θα αναφερθώ εν συντομία στην τρέχουσα κατάσταση. Αφού ο Γενικός Μηθυντής ήδη σας μίλησε το Σεπτέμβριο φέτος, παρουσιάζοντας σας αναλυτικά την τρέχουσα κατάσταση. Οπότε εγώ θα επικεντρωθώ περισσότερο στο υπόβαθρο, για να το πω έτσι. Και τέλος θα ήθελα να καλύψω εν συντομία το τι θεωρούμε ότι λειτουργήσε καλά και τι λειτουργήσε λιγότερο καλά μέχρι στιγμή σε αυτή την προγραμματική περίοδο. και όλα αυτά θα μας οδηγήσουν ομαλά και με συνοχή στην τελική ε, παρουσίαση του Διευθυντή μου για τις προτάσεις για το 2020. Η πολιτική συνοχή αποτελεί το 1 τρίτο του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Σε αυτή την προγραμματική περίοδο σχετίζεται στενά με την ε, στρατηγική Ευρώπη 2020 που βοηθά στην επίτευξη των στόχων που έχουν καθιερωθεί στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής. Όπως είπε ο Έρικ ήδη, το πραγματοποιεί αυτό επενδύοντας σε όλες τις περιοχές. Αυτό πιστεύω είναι ένας από τους βασικότερους πυλώνες της προσέγγισης της πολιτικής συνοχής. Εάν δεν έχει πολιτική συνοχή για όλε τι περιφέρειες, δεν έχει ευρωπαϊκή πολιτική συνοχή. Ε, Διότι αυτή κατεκρεματίζεται, είναι μεροληπτική και μας απομακρύνει από, την, από τα στοιχεία συνοχή και αλληλεγγύη που προσπαθούμε να πετύχουμε. Η όλη έννοια της πολιτικής συνοχής βασίζεται στην προσέγγιση εφαρμογής της, παροχής της. Βασίζεται στις βασικές έννοιες του προγραμματισμού, της εταιρική σχέσης και της κοινή διαχείρισης, της επιμερισμένης διαχείρισης. Η προσέγγιση της επιμερισμένης διαχείρισης, για να τα δούμε αντίστροφα, σημαίνει ότι η ευθύνη είναι επιμερισμένη. Επιμερισμένη μεταξύ κομισιών, κρατών μελών, περιφερειών για την παροχή της ε, πολιτικής. Αυτό γίνεται διασφαλίζοντας ε, τις ε, πιο ευρείες δυνατές εταιρικέ σχέσεις όσον αφορά την υλοποίηση των προγραμμάτων. Όπως είπαμε, αυτό είναι μια από τις βασικές αρχές του τρόπου παροχής υλοποίησης ε, της πολιτικής συνοχής. Διασφαλίζεται ότι η, η, η οικειοποίηση της πολιτικής των προγραμμάτων οργανώνεται στο πλαίσιο μιας εταιρικής σχέσης οριζόντιας ε, στη γεωγραφική περιοχή που καλύπτεται, αλλά και κατακόρυφης ε, εντός ε, της περιφέρειας του κράτους μέλους όπου απευθύνεται. Όσο το δυνατόν λοιπόν ευρύτερη εταιρική σχέση, ούτως ώστε να λαμβάνονται υπόψη όλες οι απόψεις, όλοι οι φορείς οι οποίοι μπορούν να συμμετέχουν και να συμβάλλουν στην παροχή των προγραμμάτων. Και τα προγράμματα παραμένουν ο, τα βασικά στοιχεία της πολιτικής. Ε, έχετε προγράμματα που καλύπτουν ολόκληρη την προγραμματική περίοδο με τα επιπλέον έτη που προσφέρονται για τις δαπάνε τα προγράμματα αυτά. Έτσι λοιπόν καλύπτουν συνολικά ε, μια περίοδο 9 με 10 ετών. Ένα από τα δύσκολα στοιχεία των προγραμμάτων είναι το να επιτευχθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ του ε, βαθμού λεπτομέρεια που είναι αναγκαίο για να δοθεί η κατεύθυνση προ την οποία πρέπει να κινηθεί η πολιτική, ενώ ταυτόχρονα δεν θέλουμε να είναι τόσο λεπτομερή προσπαθώντας, όταν προσπαθεί κανεί να σχεδιάσει στρατηγικά έγγραφα που καθοδηγούν τις δαπάνες για μια ολόκληρη δεκαετία. The current approach, um, in... Η σημερινή προσέγγιση στην περίοδο 14-20 καλύπτει πέντε διαφορετικά ταμεία του από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Έχουμε το Ευρωπαϊκό Αυτά ονομάζονται Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία. Όλα μαζί από κοινού. Και ένα από του βασικού σκοπού εδώ ήταν να δοθεί ένα βαθμό κοινή κατεύθυνση και συντονισμού μέσω τη χρήση μια εταιρική σχέση για κάθε κράτο μέλο, παρέχοντα ένα γενικότερο έγγραφο που αφορά την οργάνωση και δόμηση εντός κάθε κράτους μέλους όλης της διαρθρωτικής ε, χρηματοδότησης. Το άλλο στοιχείο ήταν η παροχή περισσότερων κοινών ε, διατάξεων μεταξύ των ταμείων. Ένα από τα πιο δύσκολα σημεία για τους δικαιούχους ήταν οι διαφορετικοί κανόνες που έπρεπε να ακολουθούν ανάλογα με το ταμείο στο οποίο προσπαθούσαν να έχουν πρόσβαση. Ένα από του κλάδου λοιπόν στου τομεί που προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε σε αυτή την περίοδο 14 20 ήταν να οικοδομήσουμε μια ε, κοινή προσέγγιση, όπως βλέπετε εδώ, ε, απλουστευμένες ε, επιλογές κόστους, τους κανόνες επιλεξιμότητας στα χρηματοοικονομικά μέσα. Μπορεί λοιπόν κανεί να παρέχει μια αιτιολόγηση, μια επιχειρηματολογία για να έχει πρόσβαση στα ταμεία χωρί να ασχολείται με τι επιμέρου παραλλαγέ ε, ε, των κανόνων για τα ταμεία αυτά. Πάμε στο περιεχόμενο. Η δομή για την περίοδο 14-20 βασιζόταν στους στόχους ε, της στρατηγικής ε, για το 2020 που μεταφράστηκε σε διάφορους 11 στόχους. Βλέπετε εδώ το Ευρωπαϊκό ε, Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης δραστηριοποιητικέ στους 11 στόχους, παρότι οι βασικές προτεραιότητες είναι περισσότερο οι τέσσερις πρώτες. Για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έχουμε τις προτεραιότητες 8 και 11 ουσιαστικά, που είναι πιο σημαντικές. Το δύσκολο εδώ, και νομίζω ότι ο Έρικ θα επανέλθει σε αυτό, είναι ότι υπήρξε ο κίνδυνος ε, ε, διαμερισματοποίησης, για να το πούμε έτσι, κατακαιρματισμού σε, σε ξεχωριστά πλαίσια της κάθε πολιτικής και του κάθε στόχου. Δηλαδή υπήρχε ο κίνδυνος αυτή, οι στόχοι να γίνουν κατακόρυφοι πυλώνες αδιάβλητοι και να αποτελέσουν έτσι εμπόδιο για μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση. In relation to, um, the aims and objectives. Σε σχέση με τους στόχους της πολιτικής ένας από τους βασικότερους τομείς ε, που αναπτυχθήκε σε αυτή την ανάγκη υπήρξε η ανάγκη συγκέντρωσης των επενδύσεων. Παρότι θέλουμε να υπάρχει κάποια ευελιξία ε, όσον αφορά ολόκληρο το σύνολο των θεματικών στόχων, ταυτόχρονα παρουσιάζεται και η ανάγκη διασφάλιση επαρκούς επίπεδου συγκέντρωσης ε, στις βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επικέντρωση δηλαδή στην έρευνα, της καινοτομία, στις ε, τεχνολογίες πληροφορίας και ε, τηλεπικοινωνιών, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στην μετάβαση ε, οικονομίας χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Αυτά από τον πυρήνα ε, της συγκέντρωσης για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και επίσης και στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είχαμε ενό άλλου είδους ε, ε, συγκέντρωση ώστε να διασφαλίσετε ότι τα κράτη-μέλη θα ε, πανίσουν έστω και μια ελάχιστη χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, της φτώχειας. Εκεί τίθεται το ερώτημα τη ισορροπία των ζητημάτων. Πόση ευελιξία έχει κάθε περιφέρεια να επιλέξει τι δικέ τη προτεραιότητε και πόσο ε, θα ενταχθεί σε ένα γενικότερο πλαίσιο με το οποίο πρέπει να ευθυγραμμιστεί ουσιαστικά με τις γενικότερες προτεραιότητες τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έκβαση της προγραμματικής άσκησης της περίοδου 2014-2020 έψη περιεχομένου είναι αυτό που βλέπετε τώρα στην οθόνη. Όπως βλέπετε εδώ, οι διάφοροι θεματικοί στόχοι παρουσιάζονται κατά κατηγορίες. Εδώ αν δείτε κάθε επιμέρους πρόγραμμα σε κάθε κράτος μέλος και συγκεντρώσετε, αθροίστε τις δαπάνες, αυτή είναι η κατανομή όπως το βλέπετε εδώ από το συνολικό προπολογισμό λοιπόν όπως βλέπετε περίπου 100 δισεκατομμύρια καταμεριστηκαν, επιμεριστικά στην υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων περίπου 90 δις ε, στην περιβαλλοντική προστασία και την αποτελεσματικότητα των πόρων και μια τρίτη κατηγορία περίπου 66 δις ε, στην έρευνα και καινοτομία. Ένα πράγμα που πρέπει να σχολιάσω εδώ είναι ότι ενίοτε η συζήτηση περί ευρωπαϊκής χρηματοδότησης ε, λαμβάνει τη μορφή ε, κάποια συζήτηση μεταξύ πολιτικών παραδοσιακών και νέων. Εκεί πρέπει να προσέχει πολύ κανεί τι λέει και τι λέξει επιλέγει, διότι η συνοχή μερικέ φορέ ε, περιγράφεται μια πιο παραδοσιακή πολιτική, κλασική πολιτική, παρότι εδώ βλέπετε 66 δισεκατομμύρια που έχουν επενδυθεί στην έρευνα και στην καινοτομία σε αυτή την περίοδο που διατρέχουμε τώρα κάτι που μάλλον είναι νέο παρά παραδοσιακό ή κλασικό. Ο Ερικ επίσης αναφέρθηκε στην παρουσίασή του στη σπουδαιότητα της Ιντερέγκη και της συνεργασίας, της διαπεριφερειακής συνεργασίας. Αυτό είναι ένας από τους τομείς όπου πιστεύουμε ότι η πολιτική συνοχή παρέχει πραγματική ε, προσθέμενη αξία ευρωπαϊκού επίπεδου. Η συνεργασία διασυνοριακά είναι αναπόφευκτα για την Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι που μπορεί να προσδώσει προσταμένη αξία. Αυτό είναι ένα αμφίβολο. Μέσω διαφόρων προγραμμάτων διασυνοριακών, ε, διακρατικών, διαπεριφερειακών και στην περίοδο 14-20 είδαμε αυτά τα στοιχεία σε πολλές ε, ε, γεωγραφικές περιοχές των μακροπεριφερειακών στρατηγικών. Εδώ προσθέθηκε άλλο ένα επίπεδο στρατηγικής προσέγγισης. We have indeed tried to focus more. Προσπαθήκαμε να εστιαστούμε περισσότερο πράγματι στα αποτελέσματα σε αυτή την περίοδο 2014-2020 σε σχέση με το τι κάναμε στο παρελθόν. Συχνά, και θα επανέλθουμε σε αυτό, εστιαζόμαστε στην ε, οικονομική απορρόφηση στις δαπάνες. Αλλά στην ουσία ένα από τα βασικά ερωτήματα που πρέπει να κάνουμε είναι τι έχει επιτευχθεί, όχι μόνο τι δαπανήθηκε. Οπότε γι' αυτό προσπαθούμε να αυξήσουμε τη σημασία των δικτών, της ε, υποβολής εκθέσεων, της παρακολούθησης, ούτως ώστε να προβάλλουμε, να προσφέρουμε τα αποτελέσματα όπως παρουσίασε ε, και ο Έριξ στο τέλος της παρουσίασης του προηγουμένως. Ένα νέο στοιχείο το 2014-2020 είναι αυτή η ιδέα των προϋποθέσεων για να γίνει κάποια δαπάνη. Αυτές ε, είναι γνωστές ως ρεσιμότητες εξάντε στην περίοδο 2014-2020. Το θέμα εδώ είναι να παρέχεται ένα αποτελεσματικό πλαίσιο, μια αποτελεσματική βάση για τις δαπάνες. Να υπάρχει δηλαδή να υπάρχουν κάποιε προποθέσει. Για να σα δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα, δεν αρχίζει να δαπανά χρήματα σε έργα μεταφορών, αν δεν έχει μια στρατηγική μεταφορών που θα καθοδηγεί τις δαπάνες αυτές και τον τρόπο με τον οποίο θα γίνονται. Αυτού του είδους λοιπόν οι προϋποθέσεις αποτελούν μια νέα καινοτόμο έννοια στην στρατηγική 2014-2020. Όπω είπα, θα ε, σα παρουσιάσω λίγο και την τρέχουσα κατάσταση. Εν συντομία, βεβαίω, σε αυτό το γράφημα βλέπετε την τρέχουσα κατάσταση κατά κράτη μέλο. Οι γαλαζοπράσινες ε, γραμμές δείχνουν το επίπεδο επιλογής έργων, δηλαδή η ποσότητα τη χρηματοδότησης που έχει δεσμευτεί για έργα σε κάθε κράτος μέλος και η πορτοκαλί μπάρα που είναι σαφώς χαμηλότερη είναι το ποσό χρημάτων που έχουν δαπανηθεί από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό στα κράτη-μέλη. Ο βαθμός δηλαδή εκτέλεσης είναι χαμηλότερος από ό,τι θα θέλαμε Πιστεύω ότι στο επόμενο σημείο, στην ημερήσια διάταξη θα το συζητήσει, στο, συζητώντα την απαλλαγή επιτροπή σα. Δύο μηνύματα πρέπει να υπογραμμίσουμε, πιστεύω εδώ. Το ότι παρότι ο βαθμός των δαπανών, σίγουρα ε, το ποσοστό δαπανών είναι σαφώς χαμηλότερο από ό,τι θα θέλαμε, είναι ενθαρρυντικό που βλέπουμε τα υψηλά επίπεδα δεσμεύσεων. Τι σημαίνει αυτό, ότι απόψη η υλοποίηση στα προγράμματα πράγματι προχωρούν, επιλέγονται προγράμματα και οι δαπάνε ε, γίνονται συνεπώ. Αλλά αυτό το κενό μεταξύ δεσμεύσεων και δαπανών είναι κάτι ανησυχητικό σίγουρα, τουλάχιστον για την Κομισιόν. Το δεύτερο σημείο είναι ότι αυτή είναι η πρώτη περίοδος, το 2014-2020, που μπορούμε να έχουμε στα χέρια μας τέτοιου είδους πληροφορίες. Αυτό λόγω των στοιχείων που περιλαμβάνονται στους κανονισμούς 2014-2020 ε, ε, που του έχουν συμπεριλάβει οι συνομοθέτε την υποχρέωση να αναφέρει η Κομισιόν τέτοια νούμερα, να τα συγκεντρώνει και να, να τα ε, παρουσιάζει στο Κοινοβούλιο. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο γρήγορα διδάγματα, για να το πω έτσι, που έχουμε αποκομίσει. Το θετικό είναι ότι εμείς στην Κομισιόν θεωρούμε ότι οι στενότερες σχέσεις με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο μέχρι των συστάσεων κατά χώρα έχει δώσει τη δυνατότητα στην πολιτική συνοχή να είναι πιο αποτελεσματική, αλλά και έχει δώσει και τη δυνατότητα η όλη προσέγγιση ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις πολιτικές να ε, χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη συνοχή. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα αυτών των δεσμών που έχουν δημιουργηθεί. Η εξαντέρεσιμότητα θεωρούμε ότι έχει αποδειχθεί πολύ θετική Το πλαίσιο επιδόσεων πιστεύουμε ότι αποτελεί επίση ένα θετικό βήμα για το μελλοντικό σχεδιασμό ε, της ε, αποτίμησης των αποτελεσμάτων παρότι θα έλεγα λιγότερο θετικό είναι ο τρόπος με τον οποίο ε, χαρακτηρίζουμε ε, τις επιδόσεις, ε, δημιουργώντα περισσότερο βάρος για τα κράτη-μέλη και ειδικότερα τι προγραμματικέ αρχές. Τώρα τι μπορεί να βελτιωθεί. Το έχει τονίσει ήδη πολλά έξι επιτροπή σα. Οι καθυστερήσει εκκίνηση νέων προγραμμάτων είναι από τα κρισμότερα στοιχεία τη πολιτική συνοχή. Καθυστερήσει στην αρχή μια προγραμματική περίοδου είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο να καλυφθεί αργότερα στην προγραμματική περίοδο. Ξεκινά, όταν ξεκινά μια προγραμματική περίοδος, οι καθυστερήσεις μπορούν να επηρεάσουν ολόκληρη την προγραμματική περίοδο τελικά. Παρομοίες όσον αφορά το περιεχόμενο των εγγράφων, Έχουμε την αίσθηση ότι στην περίοδο 2014-2020 ήταν πολύ μεγάλα, πολύ λεπτομερή. Χρειάζεται να ε, ακολουθούμε μια ε, πιο απλή στρατηγική. Κάτι που υποστηρίζουμε εδώ στην Κομισιόν, αλλά ίσως όχι, δεν υποστηρίζεται από άλλα όργανα, είναι ότι αυτό ο κανόνας νήσιν 3 συμβάλλει στις καθυστερήσεις στην εκτέλεση. Μειώνει την πίεση ε, για δαπάνες ε, αποτελεσματικές και γρήγορε στο πλαίσιο των προγραμμάτων. Θεωρούμε ότι συμβάλλει και αυτό ε, στις καθυστερήσεις που παρατηρούμε τώρα. Δεν θέλω να παραθέσω όλα τα προβλήματα, αλλά ευχαριστώ θα σα απαντήσω. Αλλά αυτά είναι κάποια από τα στοιχεία τα οποία έχουμε εξετάσει και τα οποία προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε καθώ μπαίνουμε στην περίοδο μετά το 2020. Ευχαριστώ. Merci Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, το περάσουμε στην περιφερειακή πολιτική για την περίοδο μετά το 2020 και προκειμένου να υπάρχει και μια κάποια συνεκτικότητα στην όλη συζήτησή μας, μπορούμε αυτή τη στιγμή να ακούσουμε τυχόν ερωτήσεις ή παρατηρήσεις. Δεν βλέπω όμως κανέναν. Πολύ ωραία. Να κάνω εγώ τότε μια παρατήρηση και στη συνέχεια να δώσω το λόγο πάλι στον πρώτο μας ομιλητή για να μας παρουσιάσει την περιφερειακή πολιτική μετά το 2020 είπατε κάτι πολύ ενδιαφέρον στην παρουσίασή σας. Όσον αφορά τη σημασία που δίδεται όλο και περισσότερο στην πολιτική συνοχή και που θεωρείται όλο και περισσότερο ως παραδοσιακή πολιτική πλέον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταλαβαίνουμε ότι θεωρείται παραδοσιακή πολιτική και λόγω της μεγάλης ιστορικής της αξίας, λόγω του έντονου παρελθόντων της. Στα πλαίσια όμως της πολιτικής συνοχής βλέπουμε ότι Υπάρχουν επιμέρους μέτρα τα οποία ανταποκρίνονται όλο και περισσότερο στις νέες προκλήσεις. Νέες προκλήσεις που θεωρούνται όλο και περισσότερο προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σας δώσω και κάποια αριθμητικά δεδομένα. Μεταξύ του 2014 και του 2020 κινητοποίησαμε πάνω από 40 δισεκατομμύρια ευρώ όσον αφορά την κλιματική αλλαγή κινητοποιήσαμε μεταξύ 2014 και 2020 πάνω από 85 δισεκατομμύρια όσον αφορά το περιβάλλον. Συνολικά λοιπόν η πολιτική συνοχής χωρίς το New Green Deal κινητοποίησε περίπου 128 δισεκατομμύρια για το περιβάλλον και για την κλιματική αλλαγή και κάτι ακόμα περισσότερο. Καταφέραμε να ανταποκριθούμε στις νέες αυτές προκλήσεις. Το ίδιο ισχύει για την κοινοτομία. Δεν γνωρίζω τα αριθμητικά δεδομένα. 65 ή 66 δισεκατομμύρια ευρώ όσον αφορά την πρόκληση της κοινοτομίας. Ναι, λοιπόν, είναι παραδοσιακή πολιτική, πολιτική συνοχής λόγω της μακράς ιστορίας της, αλλά από την άλλη μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για μια πολιτική ιδιαίτερα σύγχρονη και η οποία ανταποκρίνεται όλο και περισσότερο στις νέες προκλήσεις οι οποίες προκύπτουν και συνδυάζεται με πολλές νέες πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στη συζήτηση που κάνουμε αυτή τη στιγμή στο πλαίσιο του CFP να συνειδητοποιήσουμε ότι η πολιτική συνοχής δεν είναι απλώς μια παλιά πολιτική που σχετίζεται μόνο με την ελληνική. Προφανώς η ελληνική εξακολουθεί και αποτελεί αναπόσπαστο κεντρικό τμήμα της πολιτικής αυτής, αλλά είναι ένα μόνο τμήμα. Η πολιτική συνοχής, όπως σας είπα, αποκρίνεται και σε πολλές νέες σύγχρονες προκλήσεις. Και κάτι ακόμα, δεν μπορούμε να έχουμε πολιτική συνοχής αν η βασική αρχή της ίδιας της συνοχής δεν επιβεβαιώνεται σε όλες τις περιφέρειες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι ε, η συνοχή θα πρέπει να βιώνεται, να πραγματοποιείται και στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και στις περιφέρειες μετάβασης, αλλά και στις πιο αναπτυγμένες περιφέρειες της Ευρώπης. Συνολικά και οριζόντια θα πρέπει να εμφανίζεται αυτή η ελληλεγγύη. Και δεδομένων μάλιστα και των νέων προκλήσεων που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, τα διακυβεύματα της πολιτικής συνοχής εμφανίζονται όλο και περισσότερο στις περιφέρειες μετάβασης, αλλά ακόμα και στις πιο αναπτυγμένες περιφέρειες. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορούμε πραγματικά να καταλάβουμε την θέση της Φιλανδικής Προεδρίας, η οποία μας λέει ότι θα πρέπει να ευνοηθούν συγκεκριμένες κατηγορίες περιφερειών εις βάρος άλλων. και καταλαβαίνετε ότι το τίμημα τελικά το πληρώνουν οι περιφέρειες μετάβασης και οι πιο ανεπτυγμένε περιφέρειες οι οποίες λαμβάνουν λιγότερα κονδύλια. Κατά αυτόν τον τρόπο αποδυναμώνεται το ίδιο το σύνολο της πολιτικής συνοχή και η βασική συνιστόσα της αλληλεγγύης στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχή. Η πολιτική συνοχή μπορεί να ευοδοθεί μόνο αν πραγματικά υπάρχει συνεκτικότητα σε αυτού σε αυτές τις τρεις κατηγορίες περιφερειών. Μόνο από κοινού μπορούμε να κινηθούμε. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να έχουμε μια πολιτική συνοχή η οποία να στρέφει τη μία περιφέρεια εναντίον της άλλης και τελικά να προκαλεί ένα κατακαιρματισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έχουμε τονίσει εμείς πάρα πολλές φορές αυτό στα πλαίσια της Επιτροπής μας. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για όλες αυτές τις πληροφορίες και τις υπενθυμίσεις και σας δίνω εκ νέου το λόγο για την ε, παρουσίαση της ε, περιφερειακής πολιτικής μετά το 2020. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, για ποιο λόγο εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε μία ισχυρή πολιτικής συνοχής. Βλέπετε εδώ πέρα ένα χάρτη της Ευρώπης και βλέπετε πού βρίσκονται οι διάφορες περιφέρειες της Ευρώπης όσον αφορά το κατακεφαλήνα ΕΠΑ. Και βέβαια οι πράσινες περιφέρειες είναι οι μόνες οι οποίες βρίσκονται πάνω από τον κοινοτικό μεσόρο. Όλες οι υπόλοιπε βρίσκονται κάτω από τον ενωσιακό μεσόρο. Και ας δούμε και λίγο τα άκρα. Από τη μία πλευρά βλέπουμε το Λουξεμβούργο που έχει περίπου 260% ΑΕΠ σε σχέση με τον κοινοτικό μεσόρο και από την άλλη βλέπουμε περιφέρειες στη Βουλγαρία για παράδειγμα που έχουν κατακεφαλή ΑΕΠ κάτω από το 40% του κοινοτικού όρου. Νομίζω ότι είναι σαφές προ όλου ότι δεν μπορούμε να έχουμε μία συνεκτική ευρωπαϊκή κοινότητα με τέτοιε έντονε αποκλήσει και αντιθέσει. και αν δεν έχουν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτε τη δυνατότητα να υποφελούνται από τη συμμετοχή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνούμε λοιπόν μαζί σα ότι θα πρέπει να έχουμε μία ισχυρή πολιτική συνοχή και στο μέλλον. να αναφερθώ σε διάφορες πτυχές της πολιτικής συνοχής στις επόμενες διαφάνειες και εξ αρχή να σα πω ότι αυτό το οποίο σα παρουσιάζω είναι η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. και όπω γνωρίζετε η πρόταση αυτή επί του παρόντο αποτελεί αντικείμενο διαπραγματεύσεων ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και ορισμένε από τι προτάσει μα αυτέ έχουν ήδη τροποποιηθεί. Άρα, επομένω η διαφάνεια αυτή μπορεί να μην δείχνει την πραγματική τελική εικόνα των πραγμάτων. Παρ' όλα αυτά, ας δούμε ποια ήταν ε, τα βασικά στοιχεία που μας κίνησαν στο να δημιουργήσουμε αυτό το νέο νομικό πλαίσιο. Πρώτον, Βλέπετε στα αριστερά τη διαφάνεια ότι υπάρχουν πολλοί δικαιούχοι που έρχονται σε εμά και μας λένε: Κοιτάξτε, έχετε πολλά διαφορετικά ταμεία, πολλά διαφορετικά κονδύλια και πολλούς διαφορετικούς κανόνες. Για ποιο λόγο να μην υπάρχει ένα κοινό εγχειρίδιο κανόνων όσον αφορά τα ευρωπαϊκά αυτά κονδύλια και ταμεία. Γι' αυτό το λόγο προτείναμε αυτόν τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων που καλύπτει 7 ταμεία. Και στο πλαίσιο αυτού του κανονισμού περί κοινών διατάξεων βλέπετε κάποια βασικά στοιχεία που έχουν να κάνουν με την επίτευξη αποτελεσμάτων για όλα αυτά τα ταμεία. Είναι ατυχέ ότι δεν καταφέραμε να καλύψουμε περισσότερα ταμεία, αλλά τουλάχιστον καταφέραμε να καλύψουμε αυτά τα 7 και ήδη αυτό από μόνο το αποτελεί ένα θετικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Βλέπετε επίσης ότι τόσο για το Ταμείο Συνοχής όσο και για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακή Ανάπτυξης αλλά και για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τα παρεμφερή ταμεία έχουμε ενσωματώσει τα νομικά κείμενα στα οποία πλέον βλέπετε τις βασικές προτεραιότητες των διαφορετικών αυτών ταμείων. Για μία ακόμα φορά χρειάστηκε και εδώ να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό, για ποιο λόγο υπάρχουν τόσα πολλά διαφορετικά κείμενα και ε, χρειάστηκε να απλουστεύσουμε το όλο αυτό νομικό πλαίσιο το οποίο καθιστούσε την κατανόηση των ταμείων ιδιαίτερα δυσχερή για τους πολίτες. Γι' αυτό το λόγο συγχωνεύσαμε και ευθυγραμμίσαμε διαφορετικά τμήματα των νομικών αυτών ε, κειμένων. Και για την Ευρωπαϊκή Όμως Συνεργασία, το βλέπετε αυτό στα δεξιά της διαφάνειας, υπάρχουν κάποια καινοτόμα στοιχεία. Θα έλεγα ότι ε, η πιο επαναστατική πρόταση είναι αυτή που βλέπετε κάτω δεξιά στη διαφάνεια, το ECBM, αυτό το περιβαλλοντικό μοντέλο βασισμένο στην ε, πληροφορική και που επιτρέπει να μπορούμε να εφαρμόζουμε στοιχεία τα οποία υπάρχουν σε ένα κράτος μέλος και σε ένα άλλο κράτος μέλος συνεργαζόμενο από την άλλη πλευρά των συνόρων. Είμαστε ιδιαίτερα απογοητευμένοι που όμως ε, δεν έχει ανταποκριθεί καθόλου στην πρόταση αυτού το Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη χαιρέτησε πολύ θετικά και πολύ γρήγορα μάλιστα ενέκρινε τη θέση του, αλλά δυστυχώς μέχρι σήμερα το Συμβούλιο δεν μας έχει δώσει ξεκάθαρη θέση όσον αφορά τον διασυνοριακό αυτό μηχανισμό συνεργασίας και γι' αυτό το λόγο δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε τους τριμερείς διαλόγους και θεωρούμε ιδιαίτερα θλιβερό αυτό. Τώρα, να επιστρέψω σε αυτά που είπε ο Μόρη πριν από λίγο. Θελήσαμε να δώσουμε ένα τέλος πλέον σε αυτή την νοοτροπία κατακαιρματισμού και τομιακής μόνο προσέγγισης όσον αφορά τα κονδύλια. Επομένως, από τους 11 στόχους των ταμείων έχουμε περάσει σε 5 πλέον στόχους. Τους βλέπετε αυτού στα αριστερά της διαφάνειας. Να αναφερθώ στον τελευταίο στόχο, μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες τη. Συντοποιούμε ότι σαφώς υπάρχει ένα πρόβλημα, ότι είμαστε πολύ απομακρυσμένοι από τους πολίτε και βλέπουμε ότι ε, οι πρωτοβουλίες ε, από την βάση προς την κορυφή συνήθως είναι ιδιαίτερα επιτυχείς, γιατί καταφέρουν οι πρωτοβουλίες αυτές πραγματικά να γίνονται αποδεκτές πολύ γρήγορα και εύκολα από τους πολίτες. Ελπίζουμε λοιπόν ότι και στο μέλλον θα χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο η πρωτοβουλία αυτή προκειμένου να έχουμε καλύτερα ενστερνισμό των πολιτικών μας σε τοπικό επίπεδο. Λοιπόν, να μην σας ζαλίσω εδώ πέρα με τα διάφορα αριθμητικά δεδομένα που βλέπετε στη διαφάνεια. Αυτό το οποίο θέλουμε να πούμε με τη διαφάνεια αυτή είναι ότι δεν θέλουμε να υπάρχει μόνο μία πολύ αδύναμη κατανομή των κονδυλίων. Μας ενδιαφέρει να επικεντρωθούμε στην κοινοτομία, το κλίμα και το περιβάλλον. Αυτό ενδιαφέρει όλους ιδιαίτερως και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η εκλεγή σε πρόεδρος, ε, έχει θέσει ως βασική της προτεραιότητα το νέο αυτό σύμφωνο για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Εμείς λοιπόν πολύ σύντομα, μάλλον στις αρχές Ιανουαρίου, θα σας προτείνουμε μια νέα πρόταση για ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Δίκαιη Μετάβαση. Στόχο μα εδώ πέρα είναι να βοηθήσουμε τι περιφέρειε εκείνε οι οποίε ε, δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στους κλιματικούς μας στόχους. Θα μπορέσουμε λοιπόν μέσω του Ταμείου αυτού να υποστηρίξουμε τις περιφέρειες αυτές και μέσω της οικονομικής διαφοροποίησης αλλά θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε και τους πολίτες εκείνους οι, οποίες, οι οποίοι χάνουν τη δουλειά τους ακριβώς επειδή θα πρέπει να κλείσουν κάποιες επιχειρήσεις, για παράδειγμα βιομηχανίες εξόρυξης άνθρακα ή ενδεχομένως άλλες επιχειρήσεις να χρειαστούν να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις της κλιματικής αλλαγής. Λοιπόν, δεν θα ήθελα να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες από αυτά τα οποία βλέπετε σε αυτή τη διαφάνεια, να σταθώ μόνο σε αυτό που βλέπετε στα αριστερά της διαφάνειας, οι εξάντε ε, ερεσιμότητες είναι πολύ σημαντικές. Ε, άρχισαν να ισχύουν, θα αρχίσουν να ισχύουν μάλλον από το 2020 και πολύ συχνά βέβαια είναι μέτρα τα οποία είναι ιδιαίτερα πολύπλοκα και δεν θα πρέπει αναγκαστικά να διέπουν όλη την περίοδο προγραμματισμού. Προσπαθήσαμε λοιπόν εμείς να απλουστεύσουμε την προσέγγισή μας και να διασφαλίσουμε ότι οι ε, ενθαρρυντικέ αυτές προποθέσει όπως θα αποκαλούνται στο μέλλον, θα πρέπει να τηρούνται στο σύνολο της περίοδου προγραμματισμού. Να σας δώσω ένα-δυο ακόμα στοιχεία. Πρώτον, στα αριστερά της διαφάνειας, το δεύτερο εδάφιο, Ξέρετε ότι είχαμε μια πολύ επώδυνη εμπειρία την περίοδο που ξεκίνησε το 2014 όταν επλήγει η Ευρωπαϊκή Ένωση από την προσφυγική κρίση. Δεν είχαμε τότε καμία απολύτω δημοσιονομική ευελιξία για να καλύψουμε την κρίση αυτή μέσω των ταμείων μα. Ξέρετε ότι η ενσωμάτωση, η ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων, τα κέντρα υποδοχή, όλα αυτά θα θέλαμε το τι κάνετε, υποστηρίξουμε, αλλά δυστυχώ δεν είχαμε καθόλου χρήματα τότε. Γι' αυτό το λόγο, για την περίοδο μετά το 2020, προτείνουμε μία ενδιάμεση αναθεώρηση το 2024-2025 και θα προβλέπετε πλέον και ένα αποθεματικό ευελιξίας προκειμένου να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε πολύ πιο γρήγορα στις ενδεχόμενες μελλοντικές αναδυόμενες προκλήσεις που δεν τις γνωρίζουμε καν σήμερα. Πριν από λίγο σας είπα ότι ένα στοιχείο που μας προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία είναι αυτό που έχει να κάνει με την δυσκολία που παρουσιάζουν οι κανόνες μας. Και θεωρούμε ότι ακόμα και με τις καλύτερες δυνατές προθέσεις θα πρέπει να έχουμε κανόνες που να επιτρέπουν στους δικαιούχους μας να υποφελούνται πραγματικά από τα ταμεία μας. Γι' αυτό το λόγο προτείναμε μία σειρά δράσεων για να πετύχουμε το στόχο αυτό. Επιγραμματικά να αναφερθώ σε μία από τις δράσεις αυτές, η οποία εκ πρώτη όψεω μπορεί να μην φαίνεται πάρα πολύ σημαντική, ωστόσο ήθελα να επιστήσω σε αυτή την προσοχή σας. Τρίτο εδάφιο στα αριστερά, τεχνική στήριξη. Ξέρετε ότι ως ε, κοινοτικό δημόσιος υπάλληλο, είναι πολύ δύσκολο να δεχθώ τελικά ότι μπορεί κανείς να αποζημιωθεί για δράσεις τεχνικής αρρωγής χωρίς να δικαιολογήσει τις δαπάνες μέσω τιμολογίων. Και ακριβώς αυτό προτείνουμε εμείς τώρα. Προτείνουμε ότι θα καλύψουμε χρηματοδοτικά την τεχνική αρρωγή με βάση την εφαρμογή του προγράμματος και τίποτα παραπάνω, γιατί θεωρούμε ότι η τεχνική αρρωγή ακριβώς αυτό θα πρέπει να στοχεύει στην εφαρμογή και εκτέλεση των προγραμμάτων. 100 ευρώ για παράδειγμα μπορείτε να ζητήσετε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα πάρετε πίσω 105 ευρώ χωρίς να χρειαστεί να προσκομίσετε κανένα άλλο δικαιολογητικό. Νομίζω ότι αυτό απλουστεύει πάρα πολύ την εκτέλεση των προγραμμάτων και θεωρώ ότι προτάσει τέτοιου είδου, θα πρέπει να εφαρμοστούν και από τους συναδέλφους στα κράτη-μέλη. Ας μην αναλώσουμε τώρα πάρα πολύ χρόνο σε αυτές τις διαφάνειες που βλέπετε, γιατί ε, καλύπτουμε εδώ πέρα κάποια πολύ λεπτομεριακά ζητήματα εφαρμογής. Να επιστήσω μόνο την προσοχή σας σε ένα-δύο εδάφια της διαφάνειας αυτής. Πρώτον, Το βλέπετε στα πάνω αριστερά της διαφάνειας. Αν δούμε ότι λειτουργούν σωστά τα προγράμματα και ότι επομένω δεν υπάρχουν παρατυπίε, δεν υπάρχουν σφάλματα, τότε ουσιαστικά ω Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέμε πολύ ωραία, κανένα πρόβλημα, εμπιστευόμαστε πλήρω την Εθνική Διαχειριστική Αρχή και το σχετικό εθνικό σύστημα και ουσιαστικά δεν απαιτούμε πλέον από εσά να προσβαίνετε, να κάνετε συγκεκριμένου ελέγχου που τους ε, απαιτούσαμε συνήθως στο παρελθόν από τους δικαιούχους και τους υπόλοιπους εταίρους μας. Πρόκειται για μια γενναιόδορη προσφορά από τη δική μας την πλευρά προκειμένου να μειωθεί το διοικητικό άγχος, όσον αφορά του διαχειριστέ των προγραμμάτων, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από τι καλέ επιδόσεις του κάθε προγράμματο. Αυτό θεωρώ ότι είναι απόλυτα δικαιολογημένο και επιτρέπει σε κάθε πρόγραμμα να υποφεληθεί από τη ρήτρα αυτή, γιατί σε καμία περίπτωση δεν έχει να κάνει με το ποσό το ποσό της χρηματοδότησης, είτε πρόκειται για ένα πρόγραμμα της Ανατολικής, της Νότιας ή της Δυτικής Ευρώπης, εμείς δεν κάνουμε καμία διάκριση αρκεί το πρόγραμμα να λειτουργεί καλά. Ολοκληρώνοντας, να αναφερθώ σε ένα-δυο ακόμα ζητήματα, τα οποία μας είναι ιδιαίτερα προσφυλή. Πρώτον, τα χρηματοοικονομικά μέσα. Δυστυχώς, πάλι έχουμε εδώ πέρα την εντύπωση ότι η Φιλανδική Προεδρία το πρότεινε μάλιστα σήμερα αυτό και συζητήθηκε σε επίπεδο πρεσβευτών. Πρότεινε ακόμα μια περικοπή 7 δισεκατομμυρίων ευρώ για την πολιτική συνοχής και έχουμε την εντύπωση ότι όπως και να διαχειριστούμε την κατάσταση σε καμία περίπτωση δεν θα καταφέρουμε να φτάσουμε στα ίδια επίπεδα χρηματοδότησης που είχαμε στην τρέχουσα χρηματοδοτική περίοδο. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να είμαστε πιο αποδοτικοί, πιο αποτελεσματικοί. Και τι σημαίνει αυτό. Δεν θα πρέπει να εξαρτώμεθα μόνο από τις επιχορηγήσεις, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και εγγύσεις και δάνεια προκειμένου να καταφέρουμε να έχουμε την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη και τις ιδιωτικές επενδύσεις και κατά αυτόν τον τρόπο η δικιά μας η χρηματοδότηση να έχει μεγαλύτερο και ευρύτερο αντίκτυπο. Γι' αυτό το λόγο προτείνουμε διάφορες τροποποίησεις που είναι αρκετά μοναδικές. Για παράδειγμα, μπορεί κανείς να συνδυάσει επιδότηση με ένα δάνειο και κατά αυτόν τον τρόπο το δάνειο γίνεται πιο φτηνό ή μπορεί κανείς κατά αυτόν τον τρόπο να προσελκύσει επενδύσεις που διαφορετικά δεν θα μπορούσε να τις προσελκύσει γιατί δεν θα θεωρεί το αρκετά συμφέρον αυτό με όρους αγοράς. Επίσης, στο μέλλον θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε τις απαιτήσει ε, απέναντι στους δικαιούχους και τους διαχειριστές των προγραμμάτων όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων. Θέλουμε και εδώ να χρησιμοποιήσουμε το ηλεκτρονικό σύστημα της πολιτικής συνοχής, να έχουμε λιγότερα έγγραφα, λιγότερες γραπτές αναφορές, προκειμένου να διευκολυνθούν τα πράγματα για όλους. Τώρα, κάποια στοιχεία που έχουν να κάνουν κυρίως με χρηματοοικονομικά ζητήματα όσον αφορά τα ποσοστά κοινοτική συγχρηματοδότησης. Ε, στην τρέχουσα περίοδο έχουμε υψηλά τέτοια επίπεδα συγχρηματοδότησης, τα οποία συνδέονται με το ότι ε, ακόμα εξερχόμαστε από μία οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Υπάρχουν πολλά κράτη-μέλη που δεν είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να κινητοποιήσουν από του εθνικού προπολογισμού τα απαραίτητα ποσά τα οποία θα έρθουν να συμπληρώσουν τη δική μα τη χρηματοδότηση. Εμεί ελπίζουμε ότι από το 2021 και μετά τα πράγματα θα είναι πιο ευνοϊκά, πιο αρμονικά και γι' αυτό το λόγο προτείνουμε να μειωθεί το μερίδιο που μας συναλλογεί όσον αφορά την συγχρηματοδότηση και ελπίζουμε ότι θα το υποστηρίξουν αυτό και οι δύο συνομοθέτες, διότι καταλαβαίνετε ότι εν γέννη, μειώνοντας εμείς τη δική μας τη χρηματοδότηση, θα καταφέρουμε να αυξήσουμε το συνολικό αριθμό επενδύσεων. Όπως είπε και ο Μόρι, θέλουμε να περάσουμε στον κανόνα αποδέσμευσης ε, κονδυλίων ακολουθώντας ε, το μοντέλο 1-2. Αν δεν το πετύχουμε αυτό, τότε το όλο σύστημα λειτουργεί κατά της πολιτικής συνοχής. Υπάρχουν ε, κονδύλια τα οποία δεν εκταμιεύονται γρήγορα και δεν απορροφώνται γρήγορα, ενώ είναι διαθέσιμα. Εν κατακλείδη να σας δώσω κάποια αριθμητικά δεδομένα προκειμένου να συγκρίνουμε τον τρόπο με τον οποίο θα δοθούν τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανάμεσα στις διάφορες περιφέρειες. Βλέπετε εδώ πέρα ότι ε, ένα 75% πηγαίνει στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, που ουσιαστικά το ποσοστό αυτό παραμένει το ίδιο. Αναφέρομαι εδώ πέρα στην κατανομή των κονδυλίων, η οποία όπως βλέπετε παραμένει ίδια ανάμεσα στις δύο προγραμματικές περιόδους. Όσον αφορά τώρα αυτόν τον χάρτη επιλεξιμότητας, έχουμε τις τρεις αυτές κατηγορίες περιφερειών, λιγότερο αναπτυγμένες, περιφέρειες μετάβασης και πιο αναπτυγμένες περιφέρειες και εδώ βλέπετε τα κράτη-μέλη τα οποία θα εποφεληθούν από το Ταμείο Συνοχής, το οποίο είναι χρηματοδοτικό μέσο σε επίπεδο κρατών μελών και δεν καλύπτεται σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά όπω σα είπα σε εθνικό επίπεδο. Ολοκληρώνω στο σημείο αυτό και σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Ο λόγο στον κύριο Πεκάριαν. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. οπότε ό,τι κατάλαβα, ένας από τους βασικούς στόχους της ε, πολιτικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η βασική της αποστολή, είναι να βοηθήσει να συγκλίνουν διάφορες περιφέρειες στην Ευρώπη. Όταν ε, μελετάμε όμως τα στατιστικά της Eurostat, ε, με ευκολία βλέπουμε ότι οι διαφορές μεταξύ χωρών πράγματι συρρυκνώνονται. Μεταξύ χωρών. Όταν όμως, να, όταν όμως δούμε τα στοιχεία για τις περιφέρειες, εκεί τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Αν μετρήσουμε με βάση το περιφερειακό ε, εισόδημα, ε, θα δείτε θα δούμε ότι υπάρχουν περιφέρειες οι οποίες δεν καταφέρουν να αναπτυχθούν. Για ποιο λόγο είναι η ερώτησή μου. Μήπως θα έπρεπε να εστιάσουμε στις χώρες τις οποίες η διαφορά μεταξύ της πιο πλούσιας και της πιο φτωχής περιφέρειας είναι ε, δύο και τρεις φορές μεγαλύτερη ε, ενώ η πιο πλούσια περιφέρεια είναι δύο και τρεις φορές πιο πλούσια από την πιο φτωχή. Μήπως θα πρέπει να εστιάσουμε σε αυτές, γιατί αυτές είναι οι χώρες και οι συγκεκριμένες περιοχές οι οποίες δεν έχουν πετύχει. Υπάρχουν περιφέρειες οι οποίες έχουν ένα περιφερειακό εισόδημα, καθάριστο περιφερειακό εισόδημα, στο ίδιο επίπεδο με αυτό που είχαν πριν από δεκαετίες, ενώ όλες οι άλλες περιφέρειες έχουν γίνουν πιο πλούσιες, έχουν αναπτυχθεί. Ποιος είναι ο λόγος με τον οποίο δεν έχουμε πετύχει σε αυτές τις περιπτώσεις. Merci beaucoup. Eric Έρικ, έχεις το λόγο. Είναι πολύ σημαντικό όλα αυτά τώρα που ετοιμαζόμαστε και για την ε, Πράσινη Συμφωνία. Ε, τώρα, για το Ταμείο της Δίκαιας Μετάβασης. Πολύ καλή ιδέα. Αλλά όπως και παλιότερα, μόλις, ε, ένα, μόλις εντοπίσουμε ένα πρόβλημα, δημιουργούμε ένα καινούριο όργανο. Και δεν είναι μόνο αυτό το όργανο, είναι και άλλα όργανα και άλλα εργαλεία. Ε, αν συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση θα χειροτερεύσει η αποδοτικότητά μας, η ικανότητά μας να δρούμε αποτελεσματικά. Έτσι κι αλλιώς, τα διαρθρωτικά ταμεία λαμβάνουν υπόψη την κλιματική αλλαγή ήδη. Έχουμε αλλάξει από την παλιά δομή στην καινούργια δομή. Μετά υπάρχουν και άλλα θέματα. Πώς θα χρηματοδοτηθεί αυτό το Ταμείο τη Δίκαιης μετάβαση και πώς θα λειτουργήσει ανεξάρτητα, πώς θα έπρεπε να ενσωματωθεί στο Ταμείο συνοχή. Επίσης το σημαντικό είναι να κρατήσουμε ενωμένη την Ευρώπη και με ανησυχεί το εξή. Περιφέρειες οι οποίες δεν έχουν για παράδειγμα μετρό ή ε, μέσα μαζικής μεταφοράς. Ε, δεν δίνουν την ευκαιρία στους πολίτες τους να μην πάρουν το αυτοκίνητό τους, να μην πάρουν το αεροπλάνο κλπ. Πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Το άλλο ζήτημα που προκύπτει και από τα 13 χρόνια εμπειρίας μου είναι ότι ε, το απόθεμα επίδοσης δεν φαίνεται να διευκολύνει τα πράγματα. Το αντίθετο. Ή λοιπόν ας το καταργήσουμε ή ας το αλλάξουμε σε βάθος. και όλα αυτά θα χρειαστούν χρήματα. Οπότε καλό είναι να ξεκινήσει ένας ειλικρινής διάλογος με το Συμβούλιο. Euh, Ευχαριστούμε για αυτές τις τρεις παρουσιάσεις. Πολύ ωραία η επισκόπηση του παρελθόντος, αλλά και οι προβλέψεις για το μέλλον. η πολιτική συνοχής αναγνωρίζεται θετικά από τους πολίτες. Αν ρωτήσουμε σήμερα τους πολίτες ποια είναι τα θετικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λένε ε, ότι είναι η ενιαία εσωτερική αγορά και τα σχέδια τα οποία συγχρηματοδοτούνται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως πρέπει να είμαστε βιώσιμοι και στο μέλλον. Γιατί οι παρουσιάσεις ήταν καλές, αλλά ε, είδα μερικές αντιφάσεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι υπέρμαχος της πολιτικής συνοχής. Στα κράτη-μέλη αντίθετα υπάρχει μια πιο διχασμένη γνώμη. Υπάρχουν κάποιοι που είναι φίλοι της πολιτικής συνοχής, υπάρχει και μια ομάδα φίλων της πολιτικής συνοχής, 15-16 χώρες, αλλά κάποιες άλλες χώρες δεν είναι τόσο υπέρ ιδιαίτερα οι καθαροί χρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Σε ό,τι δεν αφορά την Κομισιόν, κάνει δηλώσεις περί μια ισχυρής πολιτικής συνοχής, αλλά ορισμένοι εκπρόσωποι γενικών διευθύνσεων επισκέπτονται τα κράτη-μέλη, κάνουν παρουσιάσεις και λένε ότι το μέλλον της πολιτικής συνοχή δεν είναι και πολύ φωτεινό. Ας ε, εστιάσουμε στα σχεδιασμένα και κεντροδιαχειριζόμενα προγράμματα. στο μέλλον θα χρειαστούμε συνδε, λύσει, συνδυασμένες λύσεις, ε, από πολλά ταμεία, ε, συμπράξεις κλπ. Ωραία. Αλλά με τους καινούριου κλιματικούς στόχους οι εταιρείε και οι περιφέρειες πρέπει να αναλάβουν δράσεις αμέσως και δεν είμαι σίγουρος ότι όλος αυτό, όλες αυτές οι συνδυασμένες λύσεις για να καλυφθούν οι μεταβάσεις, για να καλυφθεί η μετάβαση, θα έχουν χρόνο να αναπτυχθούν. Με την προστίκη νέων προτεραιοτήτων, με την προστίκη της δίκαιης μετάβασης, χωρίς περισσότερα χρήματα, δεν είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε. Θα χρειαστεί τελικά να περικόψουμε την πολιτική συνοχή για να τα καταφέρουμε. Αυτή είναι η μεγάλη, αυτές είναι οι μεγάλες μου ανησυχίες. Ελπίζω να με καθησυχάσετε με την απάντησή σας. Και μια, για ένα σχόλιο για το νησιν 3. Το νησιν τρία στις ε, υπομετάβαση περιοχές. Ε, είναι καλό διότι αυτές οι περιφέρειες χρειάζονται περισσότερο χρόνο. Οπότε το πέρασμα στο, από τον ΙΣΙΝΤΡΙΑ 3 στον 2 ελπίζω ότι θα γίνει με ένα μεταβατικό μηχανισμό ε, που θα συμβιβάζει λίγο τα συμφέροντα των διαφόρων περιφερειών. Να έχουμε δυνατότητα να ενδεχομένω κάποιε περιοχέ στον ΙΣΙΝ 3 και κάποιε στον ΙΣΙΝ 2. Ευχαριστώ. Θέλει κανείς άλλο το λόγο. Όχι, από ό,τι φαίνεται. Να προσθέσω κι εγώ κάτι δικό μου. Για την περιφερειακή πολιτική μετά το 2020. Ε, αυτή η πολιτική αποφασίζεται τώρα. Και η μάχη έχει ήδη ξεκινήσει για τον μελλοντικό ευρωπαϊκό προπολογισμό, τον μελλοντικό προπολογισμό της συνοχής. Έλεγα προηγουμένως ότι από τη μια μεριά έχουμε τις παραδοσιακές πολιτικές και από την άλλη μεριά τις νέες πολιτικές. Στην πραγματικότητα όμως θα πρέπει να βγούμε από αυτή την πόλωση. Γιατί τόσο παραδοσιακές πολιτικές όπως η πολιτική συνοχή ε, παλιότερα ήταν νέες πολιτικές. Και στην παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας υπενθυμίστηκαν τα νούμερα. Μεταξύ του 2014 και του 2020 μέσω των προγραμμάτων μας κινητοποιήσαμε 41,7 δισεκατομμύρια ευρώ για το κλίμα. 41,7 δισεκατομμύρια ευρώ για το κλίμα. Και ήμασταν οι μόνοι που έκαναν κάτι τέτοιο. 47,2 δισεκατομμύρια για το περιβάλλον. Σύνολο 120, 120 δισεκατομμύρια περιβάλλον και κλίμα. Και ακόμα δεν υπήρχε η νέα πράσινη συμφωνία στο μυαλό μας. Άρα λοιπόν η πολιτική μας είναι προσανατολισμένη προς τις νέες προκλήσεις από πιο παλιά. Έχουμε μια σύγχρονη αποδοτική πολιτική που θα γίνει ακόμα πιο αποδοτική ελπίζω στο μέλλον, που δεν είναι σε καμία περίπτωση όμως μια πολιτική του παρελθόντος ξεπερασμένη. Οπότε ο αγώνας, η μάχη την οποία δίνουμε, τα επιχειρήματα τα οποία χρησιμοποιούμε υπέρ της πολιτικής συνοχής, ε, θα πρέπει να, να ε, επικαιροποιηθούν και να επιμείνουμε σε αυτά. Η Ακούσαμε τη Φιλανδική Προεδρία σήμερα με προτάσεις για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Ε, ένα τμήμα της λύσης βρίσκεται και στην μεριά του Κοινοβουλίου και είναι εδώ ο κύριος Άλμπρεχτ ε, και θέλω να τον συγχαρώ, γενικά να συγχαρώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχει σαφή θέση υπέρ ενός ευρωπαϊκού προπολογισμού. Γιατί δεν μιλάμε μόνο για την πολιτική συνοχή. Η πρόταση της Φιλανδικής Προεδρίας είναι μια πρόταση που θάβει τι φιλοδοξίε της Ευρωπαϊκής Ένωση, ακόμα και τι φιλοδοξίε του Συμβουλίου. Και, το, και, και προφανώς και τις φιλοδοξίες της Επιτροπής Φόντερ Λάγεν. Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ πώ η καινούργια Επιτροπή θα μπορέσει με αυτόν τον προπολογισμό να ικανοποιήσει τους στόχους τους οποίους έχει θέσει. Και σίγουρα απογοητεύει το ίδιο το Κοινοβούλιο, γιατί ε, φαίνεται η Φιλανδική, ότι η Φιλανδική Προεδρία δεν βλέπει αρκετά στο μέλλον με κινητοποίηση των ιδίων πόρων που θα μπορούσε να είναι μια λύση για να εξασφαλίσουμε την απαραίτητη ισορροπία. Συζητάμε τη συναπόφαση. Συζητάμε της ε, εξουσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχει όμως ένα <laughs> Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο είναι αποφασισμένο στις δημοσιονομικές διαπραγματεύσεις να αναλάβει το ρόλο του, να αναλάβει τις ευθύνε του, γιατί πέραν της ε, πολιτικής συνοχής παίζεται, διακυβεύεται συνολικά η ευρωπαϊκή πολιτική για το μέλλον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Καθυστέρησα πολύ γιατί μόλις συζητούσαμε την τελευταία πρόταση της ε, κυρίας Βαντρελάιαν και αξιοποίησα την ευκαιρία για να πω ότι έχουμε δύο σημαντικά θέματα όσον αφορά την πολιτική συνοχή. Το ένα είναι η φιλανδική πρόταση που δεν ικανοποιεί καμία πλευρά στο Συμβούλιο. διότι δίνει λίγα παραπάνω για τη συνοχή, αλλά συνολικά αυτό που προτείνουν μπαίνει σε τρομακτικές λεπτομέρειες της πολιτικής συνοχής. Είναι πολύ ενδιαφέρον που οι πρωθυπουργοί θα συζητήσουν λεπτομέρειες για το πώς θα καθορίζονται οι δικαιούχες περιφέρειες σε συγκεκριμένα κρατημέλη. Μας έκανε μεγάλη έκπληξη αλλά είναι πολύ ε, λεπτομερές το πλαίσιο αυτό για την ε, πολιτική συνοχή. Αυτό που κάνει επί ε, εντύπωση ότι δίνουν παραπάνω χρήματα για τη συνοχή, αλλά πολύ λιγότερα για άλλου είδους ε, πολιτικές, πολιτική προστασίας και άμυνας, για παράδειγμα, κάτι που δεν βρίσκει σύμφωνες φυσικά τις υπόλοιπες χώρες, σε καμία περίπτωση. Οι αποδοκίες της Κομισιόν μας είναι ήδη γνωστοί βέβαια, αλλά εδώ τίθεται ένα πολύ επίγον ζήτημα. Πριν από μερικές ώρες η κυρία Βαντερ παρουσίασε το μηχανισμό δίκης μετάβασης ε, με κονδύλιο 100 δις. Ε, αυτό παρουσίασε σήμερα. Έγινε επίσημη παρουσίαση. Και εγώ έχω κάποια σύντομη ερώτηση προς την Κομισιόν. Πώς, ποιο ποσοστό αυτών των 100 δις θα ληφθούν από την πολιτική συνοχή, διότι το μήνυμα είναι σαφές. Το λέει ότι ένα κομμάτι από αυτά θα προέλθει από την πολιτική συνοχή. Δεν είναι ότι τα διαβάσαμε από την πολιτική συνοχή σε άλλα στοιχεία, όπω θα ανέμενε κανεί. Θα ανέμενε κανεί ότι τα κομμάτια τη πολιτική συνοχή κάποια κομμάτια της πολιτικής συνοχή θα δεσμεύονταν για το κλίμα. Θα είχαμε ήδη κάποια κονδύλια για το κλίμα, αλλά κάποια κομμάτια θα δεσμεύονταν. Δηλαδή δεν θα τα αφαιρούσαν από τη συνοχή, απλά η συνοχή θα επαναπροσανατολιζόταν στο κλίμα. Οπότε αυτή είναι η σύντομη μας ερώτηση. Ξέρετε ποιο ποσοστό αυτών των 100 δις προέρχονται από την πολιτική συνοχή. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Ολμπρέχτ, είναι σαφή η ερώτηση. Γι' αυτό ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι ήδη κινητοποιούμε πάνω από 45 δις για τον στόχο 2 και ήδη κάνουμε μια πολύ σημαντική προσπάθεια. Δίνω το λόγο στην Κομισιόν και μετά θα κλείσουμε τη συζήτηση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς δεν είμαι σε θέση να απαντήσω την ερώτηση του κ. Ολμπριχτ. Διότι θα έπρεπε να ενημερωθώ κι εγώ επαρκώς ε, θα μου φαίνονταν όμως παράξενο να κινητοποιηθούν αυτά τα κονδύλια μέσω περικοπών στον προπολογισμό για τη συνοχή. Νομίζω ότι η Κομισιόν υπήρξε πολύ σαφής και θα είναι πολύ σαφής ότι για παράδειγμα το Ταμείο Δίκαιες Μεταβάσεις που θα προτείνει η Κομισιόν θα πρέπει να ε, συμπληρώνει ε, να είναι επιπλέον της πρόταση για τον προπολογισμό και όχι να ληφθεί από εξοικονομήσεις από αλλού. Νομίζω ότι την επόμενη εβδομάδα και στο Συμβούλιο τη Ευρωπαϊκή θα εκφραστεί η Κομισιόν. Νομίζω ότι αυτό το ποσό των 100 δι είναι κάτι νέο για μένα. Δεν ξέρω ακριβώ από πού προέρχεται. Ξέρω ότι γίνονται συζητήσει με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αυτή τη στιγμή, όπου μιλάμε για ε, χρηματοδότηση ε, διαφορών ειδών, εκχωρήσεις και άλλες είδες που θα συζητηθούν. Ε, χρησιμοποιώντας και κάποιο σενάριο μόχλευσης που θα μας οδηγήσει σε αυτά τα ποσά. Ε, αυτά είναι υποθέσει όμως, δεν γνωρίζω ακριβώς, αλλά δεν νομίζω ότι θα υπάρξει μείωση του προπολογισμού τη συνοχή κατά καθιονδήποτε τρόπο. Και δεν ξέρω επίση να σα πω σε ποιο βαθμό αυτή τη στιγμή τα ποσά αυτά ήδη περιλαμβάνουν τι μελλοντικέ επενδύσει για τη συνοχή ή όχι. Για το Ταμείο Δική Μετάβαση. Δίκαιη Μετάβαση. Σίγουρα θέλουμε η πρότασή μας να είναι ευφυής. Το κατά πόσο θα εκτιμηθεί, αυτό αναμένεται να το δούμε. Αλλά αυτό που είναι προφανές, όπως έχουμε ξαναπεί, το Ταμείο Δικής Μετάβασης δεν μπορεί να αποτελέσει εργαλείο υλοποίησης της ενεργειακής μετάβασης. Διότι υπάρχουν και άλλα εργαλεία που θα συμβάλλουν σε αυτό. Όπως επίσης και τα ποσά χρηματοδότησης που είναι αναγκαία είναι τόσο υψηλά που δεν πιστεύω ότι το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης θα κατάφερνε ποτέ να ε, καλύψει αυτό το κενό, να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Εμείς πώς βλέπουμε το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης θεωρούμε ότι οι διάφορες περιφερειές δεν ξεκινούν όλες από το ίδιο σημείο. Πολλές ε, θα το θεωρούσαν εξαιρετικά δύσκολο και αυτή τη στιγμή διερευνούμε, για να σας δώσω απλά ένα παράδειγμα, την ε, Δυτική Μακεδονία στην Ελλάδα, όπου η ελληνική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να κλείσει τα ορυχεία λιγνίτη και τα σχετικά ηλεκτροπαραγωγικά εργοστάσια μέσω λιγνίτη της περιοχής, ε, κάτι που αντιστοιχεί στο 20% του ΑΕΠ νομίζω της περιοχής, χιλιάδες θέσεις εργασίας. Αυτό υποτίθεται ότι θα συμβεί μέσα στην επόμενη δεκαετία. Για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να δώσεις μια νέα προοπτική και ένα νέο οικονομικό μοντέλο στην περιοχή αυτή. για να δημιουργηθούν στο μέλλον οικονομικές δραστηριότητες και θέσεις εργασία. Πώς το βλέπουμε εμεί λοιπόν. Ε, θεωρούμε ότι το Ταμείο Δίκαιη μετάβαση θα συνοδεύει, θα παράλληλα με αυτή τη μετάβαση. Θα βοηθήσει ανθρώπους που θα βρεθούν άνεργοι να βρουν νέε δουλειές ή όπως είπα να υποστηρίξουν νέες ε, οικονομικές δραστηριότητες μικρομεσαίε επιχειρήσει ή άλλου είδου εταιρείε για να καλύψει αυτές τις ζημίες και απώλειε. Αλλά δεν θεωρούμε ότι το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης θα χρηματοδοτήσει αυτό καθ' αυτό την ενεργειακή και κλιματική μετάβαση. Έχουμε άλλα εργαλεία για αυτό το σκοπό. Τώρα επιστρέφοντας ε, στον κανόνα ε, νήσιν 3, νήσιν 2, για μα. αυτό που έχει σημασία είναι ότι στο τέλος τη επόμενη προγραμματικής περίοδου θα πρέπει να έχουμε συν δύο. Πώς θα το καταφέρουμε, αυτό απομένει να συζητηθεί. Μπορούμε να βρούμε όλοι μαζί με έναν τρόπο αποδεκτό για όλους. Αλλά θέλουμε να επιστρέψουμε στο συν δύο. Και να σας υπενθυμίσω ότι στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο είχαμε νη συν δύο. Και ουσιαστικά κανεί δεν είπε ότι αυτό έχει παρουσιάσει πρόβλημα. Στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο έχουμε χαλαρώσει τον κανόνα αυτών. Έχουμε ίσως αλλάξει κάπως και το σύστημα παραδοσή μα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν νέοι κανόνε που οδήγησαν προφανώ σε κάποιε καθυστερήσει, αλλά αυτή η δικαιολογία δεν ε, θα ε, υπάρχει πια στο μέλλον, γιατί δεν πρόκειται να αλλάξουμε κάτι άλλο, απλά θα πλουστεύσουμε τα πράγματα. Θα μειώσουμε τι διαδικασίε, όλα τα διαδικαστικά, οπότε δεν υπάρχει δικαιολογία για να πούμε ότι χρειαζόμαστε παραπάνω χρόνο για να προσαρμοστούμε στους κανόνες. Δεν θα υπάρξουν νέοι κανόνες, απλά κόψαμε κάποιους κανόνες. Οπότε δεν αιτιολογείται η παραμονή στο νησιν 3 για ολόκληρη την προγραμματική περίοδο μετά το 2020 και τέλος συμφωνώ απόλυτα που είπε η αυτό που μα ανησυχεί περισσότερο, όλο και περισσότερο, είναι ότι οι διαφορέ και οι ανισότητε εντό των κρατών μελών αυξάνονται και εντείνονται. Το παρατηρούμε σχεδόν παντού. Υπάρχουν κάποιες ε, περιοχές μεγαλοπόλεων, για να το πω έτσι, ε, που σημειώνουν ταχύ ανάπτυξη. Εκεί υπάρχει η καινοτομία, τα πανεπιστήμια, οι επιχειρήσει, επιχειρήσεις, startup, ε, η επίδραση όλων των οικονομικών αλληλεπιδράσεων εκεί, όλες οι νέες θέσεις που έχουν δημιουργηθεί εκεί και μετά βλέπουμε άλλα μέρη σε κάποιες χώρες, γεωργικά ως επιτοπλίστων, αγροτικά ως επιτοπλίστων που μένουν πίσω και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Ευρώπη, συμβαίνει παντού στον κόσμο και το ερώτημα που τίθεται είναι τι μπορείς να κάνεις, τι μπορεί να κάνει κανείς για να μετριάσει αν είναι τι άλλο το πρόβλημα αυτό, διότι η επιλογή του να πει, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε με την υπόλοιπη χώρα οπότε απλά την αφήνουμε πίσω δεν είναι λύση, δεν λειτουργούν έτσι τα πράγματα βλέπετε ήδη πώ είναι οι κίνδυνοι και πώ εκδηλώνονται σε κάποιε ε, συμπεριφορές ψηφοφόρων σε κάποια κράτη-μέλη αρκεί να κοιτάξετε γύρω σα. Μιλάμε για πολίτε οι οποίοι αισθανόνται ότι του έχουμε αφήσει πίσω, ότι κανεί δεν ενδιαφέρεται για αυτού και οι οποίοι δεν φαίνεται να θεωρούν ότι έχουν μέλλον. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε αυτό απλά να συμβαίνει και να επικεντρωθούμε σε κάποιου πόλου ανάπτυξη που έχουμε που είναι ελάχιστοι. Πρέπει να βρούμε λύσει και για τις, τα υπόλοιπα μέρη τη κάθε χώρα. Αλλά δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε μόνο το πολιτική συνοχή. Ο προπολογισμό τη είναι υπερβολικά μικρό, ανεπαρκή για να κάνει διαφορά σε πολλά μέρη. Όπω είπα, μπορούμε να παρέχουμε κίνητρα, να παρέχουμε υποστήριξη, αλλά σε τελική ανάλυση χρειάζονται πολλά περισσότερα. Δεν μπορούμε να αναμένουμε λύσεις για κάθε πρόβλημα από την πολιτική συνοχή. Σε ευχαριστώ. Δύο γρήγορες απαντήσεις ε, βάσει κάποιων ερωτήσεων που έγιναν από τον κύριο Μπέρκβιστ, αν δεν κάνω λάθος. Εξέφρασε αμφιβολίες όσον αφορά το αποθεματικό επιδόσεων. Πώ λειτουργήσε από το 2014 μέχρι το 2020. Δεν μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε. Και εμείς κοιτάξαμε την ίδια κατάσταση, τις δυσκολίες, τις προκλήσεις, το επιπλέον άχθος ε, σε αυτή την περίοδο και τα συγκρίναμε αυτά με τα... κάναμε μια αντιπαραβολή με τα ωφέλη που ενδεχομένως παρέχει και γι' αυτό το λόγο μεταξύ άλλων προτείνουμε να μην συνεχιστεί στην περίοδο μετά το 2020 ενδείξεις ε, μας λένε ότι και οι δύο συνομοθέτε συμφωνούν με αυτή την προσέγγιση. Είναι ένα καλό παράδειγμα θετικού διδάγματος ε, που θα μα οδηγήσει να βελτιώσουμε κάτι από την μια περίοδο στην επόμενη. Το επόμενο σημείο σχετίζεται με περιοχές με πιο περιορισμένες μεταφορές, ε, δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κάποιε περιοχέ, Δείτε τις Αζόρες για παράδειγμα ως παράδειγμα. Δεν είναι παρά ένα παράδειγμα Βάσει παλαιότερης εμπειρίας δεν έχουμε πιστεί κατά πόσο προσφέρει κάποια αξία το να υποστηρίζουμε ε, υποδομές αεροδρομίων με την πολιτική συνοχή. Αυτή είναι μια από τι εξαιρέσει που έχει συμπεριλάβει η Κομισιόν στι προτάσει τη. Αλλά χρειαζόμαστε μια ιδιαίτερη εξαίρεση για τις εξόχως ε, απομακρυσμένε περιοχές δεδομένη τη γεωγραφική του κατάσταση, θέση των ιδιαίτερων δυσκολιών όσον αφορά τι μεταφορές. Ε, χρειάζεται εκεί μια απόκριση όσον αφορά τι περιοχές αυτές. Οπότε εδώ βλέπετε ένα παράδειγμα, ελπίζω, του πόσο προσαρμόστε στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο η πολιτική συνοχή και η περιφερειακή πολιτική. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθεί να πρέπει να προσαρμόζεται στι ιδιαίτερε συνθήκε μια ε, περιοχή και ιδιαίτερα των εξόχων από μακρισμένων περιοχών. Ευχαριστούμε. Πριν κλείσουμε τη συζήτηση, θα δώσω το λόγο στον Αντρέι Νοβακόφ. Ευχαριστώ πολύ. αν η πρόεδρος Φοντελάιεν ε, ανακοίνωσε πριν από μισή ώρα έναν μηχανισμό μετάβασης, ε, τότε θα πρέπει να γίνουν και απαραίτητε ε, τροποποίησεις στον CPR. Θα κάνετε εσείς τις αλλαγές αυτές, είναι έτοιμες, αν όχι πότε θα παρουσιαστούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, Ακούσαμε τις παρατηρήσεις από τους εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αποτολμήστε να κάνετε και κάποιες ε, ανακοινώσεις. Θα εμβαθύνουμε στην ε, συζήτηση αυτή με την ε, πολιτική συζήτηση που θα διεξάγουμε με την αρμόδια επίτροπο, η οποία πολύ σύντομα θα έρθει στην Επιτροπή μας. Σε κάθε περίπτωση, σας ευχαριστώ για την παρουσίαση των μελετών αυτών. Ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες και όπως είδατε οδήγησαν σε πολύ επικοδομητικές συζητήσεις, οι οποίες μας επέτρεψαν επίσης να ξαναθυμηθούμε τα πιο θεμελιώδη στοιχεία της πολιτικής συνοχής. Σας ευχαριστούμε πολύ και περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, που έχει να κάνει με την γενική απαλλαγή όσον αφορά τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2018. Η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού είναι η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή. Η δική μας συντάκτρια γνωμοδότησης, η κυρία Κουντατζάρ, είναι παρούσα και θα μας κάνει μία παρουσίαση του σχεδίου γνωμοδότησής της. Σας υπενθυμίζω ότι η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης τροπολογιών είναι η Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου στις 6 ώρα το απόγευμα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μετά την ανταλλαγή απόψεων που είχαμε στις αρχές Νοεμβρίου, θα ήθελα να σας τονίσω τα σημαντικότερα στοιχεία τα οποία αποφάσισα να συμπεριλάβω σε αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης. Το μάλλον ο περιορισμό των 1500 λέξεων δεν μου επιτρέπει να συμπεριλάβω όλα τα στοιχεία τα οποία θα ήθελα να συμπεριλάβω σε αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης. Λέω πάντως ότι υπάρχει μια γενικότερη θετική τάση μειώνεται το ποσοστό σφάλματος τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. Το ελεγκτικό συνέδριο για την πολιτική, οικονομική, κοινωνική και δαφική συνοχή θεωρεί ότι το ποσοστό σφάλματος είναι 5%, υψηλότερο δηλαδή από ό,τι ήταν για τον προπολογισμό του 2017. Τότε είχαμε ποσοστό σφάλματος 3% και λίγο υψηλότερο για τον προπολογισμό του 2016. Τότε ήταν γύρω στο 4%. Στο σχέδιο γνωμοδότησής μου λέω επίσης ότι δεν θα πρέπει να θεωρούμε ότι η ύπαρξη σφάλματος σημαίνει και ύπαρξη απάτης. Τούτο λεχθέντον βέβαια θα πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας την κατάσταση αυτή, γιατί σε αυτή την πολιτική έχουμε δει ότι τουλάχιστον για το 2018 το ποσοστό σφάλματος ήταν πάνω από τον ενωσιακό μεσόρο. Όπως σας είπα πριν από ένα μήνα, θα μπορούσε να σημειωθεί πρόοδος κυρίως στο 44% των μη επιλέξιμων δαπανών. Έχουμε επίση κάποιε παραβάσει των κανόνων τη εσωτερική αγορά, γύρω στο 40% και έλλειψη αποδεκτικών εγγράφων, 11%. Όπως μας υπενθύμισε ο Κρίστιαν Γκέρ στην ανταλλαγή απόψεων που είχαμε, Μερικές φορές υπάρχει γενικότερη τάση από τα κράτη-μέλη να υπεριθμίζουν κάποιες πτυχές της πολιτικής συνοχής, ιδίω το ζήτημα των τομέα της εφαρμογής. Αυτό το τονίζει και το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο στην έκθεσή του. Έτσι λοιπόν, δεν μπορώ παρά να πω ότι θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω απλουστεύσεις στη διαδικασία μετά το 2020. Τα αναφέρω όλα αυτά στο σχέδιο γνωμοδότησης που σας υποβάλλω σήμερα. Απλούστευτοι κανόνε επιλεξιμότητα ενδεχομένω να οδηγήσουν και σε χαμηλότερα ποσοστά σφάλματο. Επίση, στο σχέδιο γνωμοδότησή μου τονίζω και ένα ακόμα σημαντικό ζήτημα. Η απορρόφηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, η οποία εξακολουθεί να είναι βραδύτερη από ό,τι είχε προγραμματιστεί. Έως το τέλος του 2018 μόνο 27,3% των κονδυλίων αυτών είχε απορροφηθεί θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα βαθύτερα αίτια της χαμηλής αυτής απορρόφησης, όχι μόνο στα πλαίσια της διαδικασίας απαλλαγής, αλλά πιο σημαντικά παρακολουθώντας πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Μολονότι έχει εκφραστεί, έχουν εκφραστεί πολλές αποδοκιμασίες όσον αφορά τον λεγόμενο κανόνα 1 3, θεωρώ ότι ε, στα πλαίσια της επόμενης περίοδου προγραμματισμού θα πρέπει να αποφύγουμε τα λάθη που είχαν γίνει στο παρελθόν και είχαν οδηγήσει σε χαμηλά επίπεδα απορρόφησης. Ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα αναλάβουν τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη της καθυστερημένης εφαρμογής των ΕΔΕΤ και των επιπτώσεων που είχε αυτό. Θα πρέπει το ευρωπαϊκό, το εθνικό και το τοπικό επίπεδο να συνεργαστούν περισσότερο, προκειμένου να διασφαλίσουμε υψηλότερα επίπεδα απορρόφησης στο μέλλον. Δεν μπορώ στο σχέδιο αυτογνωμοδότησης λόγω του περιορισμού των λέξεων να φέρω δύο ακόμα ζητήματα πολύ σημαντικά όμω. Το έργο των εθνικών ελεκτικών αρχών και το ότι θα πρέπει να έχουμε πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά συστήματα επιδόσεων όσον αφορά το πρώτο ζήτημα, τις εθνικές ελεκτικές αρχές. Μολονότι έχουν εφαρμοστεί πολλέ βέλτιστες πρακτικέ, θα πρέπει να γίνουν ακόμα περαιτέρω βελτιώσει προκειμένου να παρακολουθείτε σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο καλύτερα η διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων. Θα πρέπει να έχουμε δείκτε επιδόσεων. Αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική προκειμένου να αξιολογούμε πραγματικά τα επιτεύγματα τη πολιτική συνοχή. Χρειαζόμαστε δείκτε οι οποίοι θα μα δίνουν τι σωστέ, ακριβεί πληροφορίε, πληροφορίε και δεδομένα υψηλού ποιοτικού επίπεδου. Μόνο βάσει των δεδομένων μπορούμε να πάρουμε σωστέ αποφάσει. Σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα και προσβλέπω στι παρατηρήσει σα και θα συζητήσουμε βέβαια και τις ε, τροπολογίες που ενδεχομένω να καταθέσετε μέσα σε επόμενες ημέρες. Σας ευχαριστούμε πολύ για την λεπτομεριακή αυτή παρουσίασή σας. Να δώσουμε τώρα το λόγο στους ασκιώδεις εισηγητές, ο κύριος Τάμας Ντόιτς, εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος πρώτος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συναδελφοί. Eh, Ευχαριστώ πολύ για αυτή τη ε, δουλειά. Η εισήγησή σα στο προσχέδιο αυτό είναι πολύ καλό. Όπως, είπε και η, όπως είπατε εσείς ως εισηγήτρια, ε, Υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν μπορέσαμε να συμπεριλάβουμε γιατί είχαμε περιορισμό προ τον όγκο, των αριθμών των λέξεων. Όμω θα πρέπει να αναφέρουμε τρία σημαντικά θέματα. Πρώτον, την απλοποίηση. Το είπε και η Κομισιόν στην παρουσίασή της, το παρουσίασε πολύ ξεκάθαρα. Είναι κάτι πολύ θετικό πρέπει να αποτελεί κοινή πρόθεση. Δυστυχώς όμως προχωράει πολύ αργά. Όλο μιλάμε για απλοποίηση, αλλά όλο και, περισσότερο, όλο και περισσότερες περίπλοκες διαδικασίες εισάγουμε στο σύστημα. Οι δικαιούχοι οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, οι διαχειριστές των σχεδίων δεν ξέρουν τι να κάνουν για να διαχειριστούν όλους αυτούς τους κανόνες που υπάρχουν. Το ερώτημα πραγματικά τίθεται αν η Κομισιόν θα καταφέρει να απλοποιήσει το σύστημα. Η Κομισιόν μιλάει συνεχώ για απλοποίησει, αλλά οι προτάσει είναι όλο και πιο περίπλοκε. Το ίδιο και το Συμβούλιο. Και εμεί μιλάμε συνεχώ για απλοποίηση. Τι θα κάνουμε. Δεύτερον, η χαμηλή ταχύτητα, οι, οι αργοπορίες που εμφανίζονται στα σχέδια, στην εφαρμογή σε 7 χρόνια φοβάμαι ότι θα βρισκόμαστε στην ίδια ακριβώς κατάσταση. Ίσως δεν θα είμαστε εμείς αυτήν την αίθουσα. Αλλά και πάλι θα είμαστε καθυστερημένοι σε σχέση με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Τι σημαίνει τώρα, αργεί, καθυστερεί ο προγραμματισμός, ξεκινάνε καθυστερημένα τα σχέδια, καθυστερούν στην εφαρμογή τους ακόμα περισσότερο και μετά συσσωρεύουμε καθυστερήσεις τις οποίες δεν μπορούμε μετά ε, αργότερα να απορροφήσουμε. Δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι, έτσι. Δεν είναι δική μας ευθύνη αλλά θα ξεκινήσει η νέα προγραμματική περίοδος, πάλι καθυστερημένα, σε μερικούς μήνες. Ειλικρινά δεν ξέρω τι θα γίνει σε 7 χρόνια. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξο. Ζητείτε ελαστικότητα, ζητάμε μάλλον να είναι πιο ελαστικά τα τα χρηματοδοτικά όργανα και τα προγράμματα και οι κανόνες, αλλά οι πρώτες φιλανδικής προεδρίας είναι ακόμα πιο γραφειοκρατική και πιο αυστηρή. Ο Γιάννη έχει εμπειρία με το πολιτές μεσονομικό πλαίσιο Ίσως ε, θα πρέπει να είμαστε πιο ριζοσπαστική, να, Δηλαδή, να δώσουμε βάρος στις διαπραγματεύσεις, στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα πρέπει να αγωνιστούμε για να αυξηθεί η απλοποίηση, να, να γίνει μια πραγματική απλοποίηση, ε, γιατί αλλιώς δεν θα τα καταφέρουμε. Merci beaucoup. Ευχαριστούμε πολύ για την ομάδα Renew. Κανονικά είναι ο Κριστιαν Κίνα, ο οποίος είναι σκιώδη. αλλά έμαθα ότι απουσιάζει. Ο κύριο Κότεκ θα παρουσιάσει για την ομάδα Renew. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους του σκιώδου συζητητής μας ε, για λόγους εκτέκτης ανάγκη. Ε, δεν μπόρεσε να βρίσκεται εδώ αλλά θα σας παρουσιάσω εν συντομή τη θέση του. Ο κύριος Κινέα καλωσορίζει και ευχαριστεί την κυρία Κουταγιάρα για τη γνωμοδότηση αυτή. Είναι εξαιρετική. Επισημαίνει την αύξηση του συντελεστή σφάλματος για την πολιτική συνοχή από 3 σε 5% για το 2018. Βάσει της εκθέσης της ΕΚΑ σημειώνονται δύο πραγμάτα. Η απλούστευση που υποστηρίζει και η κυρία Κουτέα και ο κύριος Ντόιτς τα είπαν οπότε θα τα αναλύσω αυτό. Το δεύτερο σημείο είναι η παράτυπη παρακράτηση πληρωμών από διάφορες διοικητικές αρχές ε, από τους δικαιούχους που εξακολουθεί να υπάρχει ως πρακτική. Εδώ πιστεύει ο Σκιώδης ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποια ειδική έκθεση για την σύνδεση μεταξύ των καθυστερούμενων πληρωμών και της ποιότητας των αποτελεσμάτων και θα πρέπει να ε, εξεταστεί αυτό το φαινόμενο αδικαιολόγητης καθυστέρησης πληρωμών προς τους δικαιούχους. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν βλέπω το συναδελφορό να είναι εδώ. Οι πράσινοι θα μας στείλουν γραπτός τη θέση τους. Το ίδιο και ο Ραφαέλε Φίτο και η Μαρτίνα Μιτσέλ που μου φαίνεται λείπει επίσης. Πριν δώσω το λόγο ξανά στον εισηγητή μας. Στην εισηγήτρια παρακαλώ, θα κάνω κάποια σχόλια, έχετε απόλυτο δίκιο όσον αφορά την απλούστευση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το 2014 οι δικαιούχοι κληρονόμησαν μια αλλαγή συστήματος, σχεδόν μια επανάσταση του ζητήθηκε. Και αυτό δεν βοήθησε καθόλου στην απορρόφηση των κονδυλίων. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και στο ρόλο μας ως νομοθέτες. Για τη νέα περίοδο λοιπόν που ξεκινά, εμείς προσδοκούσαμε από την Κομισιόν κανονισμούς που δεν θα ε, φέρουν τα πάνω κάτω στο σύστημα και εμεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μερικέ φορέ δεν ενδέχνουμε απόλυτη συνοχή σε σχέση με αυτού του ε, στόχου. Έχουμε και εμεί τα δικά μα προβλήματα ω συνομοθέτε. Ε, οπότε εδώ και εκεί κάπου περιπλέκουμε τα πράγματα. Οπότε ελπίζω ότι στους τριλόγους θα καταφέρουμε να επιλύσουμε και να ξεφορτωθούμε ότι είναι περιττό και να παραμείνουμε σε προγράμματα τα οποία θα είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, πιο ε, εύκολα στη χρήση για όλο τον κόσμο στην Ευρώπη. Δίνω το λόγο στην εισηγήτρια, αν θέλει να ξαναπάρει το λόγο. Πολύ σωστά αυτά που λέτε και εγώ αναμένω τα γραπτά σχόλια των σκιωδών που δεν ήταν παρόντα σήμερα. Η απλούστευση πράγματι είναι πολύ σημαντική. Τονίζω και ξανά πόσο σημαντικό είναι να συνεχίσει τις εργασίες της η Επιτροπή ε, Ρέτζι, ε, υποστηρίζοντας περισσότερη απλούστευση για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να λάβουμε υπόψη του σημερινού κανόνε και να δούμε πω είναι ο καλύτερο τρόπο να του τροποποιήσουμε με αυτό υπόψη μα. Είναι θέμα και διοικητικών ικανοτήτων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν ε, στα θέματα αυτά. Αναμένω να δούμε τη συνέχεια τη διαδικασία και τη μελλοντική μα συνεργασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να κάνει μια παρατήρηση. Thank you, Mr. Chair. Just perhaps... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο-τρεις παρατηρήσεις έτσι στα γρήγορα. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια πρώτα απ' όλα για τη διορατικότητά της. Δεν διαφωνούμε σε πολλά. Επίσης λυπούμεθα που ο συντελεστής φάλματος αυξήθηκε από το ένα έτος στο επόμενο παρότι θέλω να τονίσω ότι είναι σαφώς μικρότερος από ό,τι υπήρξε στο παρελθόν. Κάτι άλλο για την απλούστευση. Όπως τόνισε και ο διευθυντής μου στο προηγούμενο με τις διαταξής, αυτό υπήρξε ένας από τους βασικότερους σκοπούς ε, της Κομισιόν το προσπάθησε να το ενσωματώσει στην περίοδο μετά το 2020 η Κομισιόν. Ένα σημείο συγκεκριμένα προσπάθησαμε να εξετάσουμε σε θέματα απλούστευση. Συχνά γίνονται συζητήσει περί απλούστευση. κάτι που συχνά οδηγεί σε αλλαγέ. Ε, σε μια απόπειρα απλούστευση των πραγματών, όταν αλλάζει όμως μια υπάρχουσα προσέγγιση, έναν υπάρχοντα κανόνα, δημιουργεί ένα νέο σύστημα το οποίο κάποιο πρέπει να μάθει. Κάποια από τα στοιχεία λοιπόν στα οποία προσπαθούμε να εστιαστούμε για την περίοδο μετά το 2020 είναι τι μπορούμε να εξαλείψουμε τελείω. Γιατί όταν εξαλείφει κάτι τελείω, εξαλείφει την ανάγκη του να μάθει κανεί κάτι καινούριο και απλουστεύει τη διαδικασία σημαντικά. Αυτό κάναμε εμεί στον ορισμό των αρχών, στο σύστημα ελέγχου της διαχείρισης ε, θα ε, εξαλειφθεί στην επόμενη περίοδο τα σχόλια του κ. Ντόιτ για τον κίνδυνο να βρεθούμε στην ίδια κατάσταση, να παραμείνουμε στην ίδια κατάσταση και για, 7 χρόνια. Αντιλαμβάνομαι αυτό που λέει και ελπίζω να είναι λάθος αυτό που λέει και ελπίζω να μην τον εκνευρίζω που το λέω αυτό. Κάποια από τα πράγματα που εξετάζουμε στην αρχή της περίοδου, την άρση του διορισμού των αρχών συντομότερα, σαφέστερα έγγραφα, σημαίνει ότι η αρχή της προγραμματικής περίοδου θα χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη ταχύτητα και όπως είπα όσο πιο ταχύς είσαι στην αρχή τόσο πιο έγκαιρα προλαβαίνεις να τα καταφέρεις. Η καθυστερή στην αρχή πιστεύω ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα στην πολιτική συνοχή. Είμαστε αισιόδοξοι λοιπόν ότι αυτά που έχουμε προτείνει θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά. Ευχαριστώ. Merci Ευχαριστούμε πολύ. Σας υπενθυμίζω ότι η καταλεκτική ημερομηνία κατάθεσης τροπολογιών είναι η Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου, 6 ώρα το απόγευμα. Ευχαριστούμε τη συντάκτρια τη Γνωμοδότηση και όλους τους συναδέλφους οι οποίοι εμπλούτησαν με τις παρεμβάσει του στη συζήτηση. Νομίζω ότι ε, φτάσαμε έτσι ε, στο τέλος της σημερινής μας συνεδρίασης. όσοι δεν προβλέπετε να συμμετάσχουν στην συνεδρία των τονιστών, καλούνται να αποχωρήσουν από την αίθουσα γρήγορα και χωρίς να κάνουν θόρυβο. Σας ευχαριστώ πολύ. Je rappelle cependant que nous nous retrouverons demain ότι θα συνδράσουμε βέβαια πάλι αύριο το πρωί στις 9 η ώρα θα ξεκινήσουμε με ψηφοφορίες όσον αφορά το Euroforum και όσον αφορά τα υπόλοιπα σημεία της ημερήσιας διάταξης.